Meine sehr verehrten Damen und Herren, Λοιπόν, σας καλωσορίζω αγαπητοί συνάδελφοι στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, την οποία οπωσδήποτε έχετε στην διάθεσή σας. Συμφωνείτε. Εμένα δεν μου έχει ζητήσει κανείς κάποια αλλαγή, οπότε εγκρίνεται υποθέτω. Να σας υπενθυμίσω επίσης πως είναι δημόσια η συνεδρίασή μας με την έννοια ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε επίσης ε, και τους διερμηνείς και να περάσουμε στην έγκριση των πρακτικών της ε, Δευτέρας, 5ης, 16ης και 17ης Δεκεμβρίου. Έχετε κάποια παρατήρηση? Όχι. Οπότε εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το υπαριθμόν 4 διαδικασία απαλλαγής, Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεχίζουμε με τους ε, επιτρόπους. Ο αρμόδιος ηγητής είναι ο Μάρκους Πίπερ, τον οποίο βεβαίω καλωσορίζω και βεβαίω καλωσορίζω και τον κύριο Επίτροπο, τον κύριο Άντορ. καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μα. Περνάμε λοιπόν αμέσω στην ημερήσια διάταξη. Θα δώσω λόγο λοιπόν στον εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρακαλώ. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μέλη της Επιτροπής, εξ ονόματος του Ελληνικού Συνεδρίου είναι τιμή μου να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα του κεφαλαίου 6 της ετήσιας έκθεσης του 2012 για το θέμα της απασχόλησης και των κοινωνικών ζητημάτων. Το 2012 το Ελληνικό Συνέδριο ε, έκανε για δεύτερη φορά μια συγκεκριμένη αξιολόγηση για τα ζητήματα απασχόλησης ε, και κοινωνικών υποθέσεων. Έτσι θα μπορέσουμε καλύτερα να δούμε τα ζητήματα που αφορούν την απασχόληση και τα κοινωνικά που μια φορά διαφέρουν από αυτά τα οποία είναι στο κεφάλαιο 5, δηλαδή περιφερειακή πολιτική, μεταφορές και ενέργεια. Οι δαπάνε της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν σε αυτόν τον τομέα ήταν 13,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012. Ήταν δηλαδή μια αύξηση 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι 96% των δαπανών. Ως τμήμα των δαπανών συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι υπό τον κοινό έλεγχο της Κομισιόν και των κρατών μελών και υπόκειται στους ίδιους κανόνες όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Ο βασικός κίνδυνος για την ομότητα και την κανονικότητα των ε, δαπανών βεβαίως προκύπτει από την άειλη φύση των δαπανών σε ανθρώπινο κεφάλαιο, την ε, ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων και τους πολλούς και μικρούς εταίρους που εμπλέκονται στην εφαρμογή των έργων. Οι αυτοί οι παράγοντες προσφέρονται για μη συμμόρφωση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες επιλεξιμότητας και καταλήγουμε σε μη επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες δεν ανοιχνεύονται ή δεν διορθώνονται από τα συστήματα ελέγχου που υπάρχουν είτε στο επίπεδο κράτους μέλους είτε στο επίπεδο κομισιών. Το συνέδριο έλεγξε ένα δείγμα 180 συναλλαγών που ήταν κυρίως ενδιάμεσες τελικές πληρωμές σε έργα που πλήρωσε η Κομισιόν το 2012 το ελεγκτικό συνέδριο έλεγξε το κατά πόσον είχαν ε, συμμορφωθεί αυτές οι πληρωμές με τους υφιστάμενους κανόνες συνολικά. Λοιπόν, τα ευρήματά μας δεν άλλαξαν πολύ από τα προηγούμενα έτη. Καταλήξαμε πως το ποσοστό σφάλματος ήταν μεταξύ 1,3 και 5,1% και το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος ήταν 3,2% ενώ το 2011 ήταν 2,2% όπως τονίζει το συνέδριο, σφάλμα δεν σημαίνει οπωσδήποτε απάτη ή σπατάλη. Η συχνότητα σφάλματος μειώθηκε από 40% στο 35% το 2012 και 63 από τις 180 συναλλαγές είχαν κάποια σφάλματα. Όσον αφορά το κεφάλαιο 5, για πάνω από τις μισές ε, από τις ε, συναλλαγές που είχαν οποιοδήποτε είδος λάθους, δηλαδή 67% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες στην διάθεση των αρχών των κρατών μελών και θα μπορούσαν να είχαν ανοιχνεύσει και διορθώσει κάποια προβλήματα πριν βεβαιωθούν οι δαπάνες προς την Κομισιόν. Έτσι, μία πρόσφατη έκθεση ελέγχου από την Γενική Διευθύνση Απασχόλησης που ε, αφορά των της ελέγχους ε, πρώτου βαθμού επιβεβαιώνει ακριβώς τις αδυναμίες αυτές. Το 2012 το κεφάλαιο 6 εμβαθύνει στην ανάλυση των σφαλμάτων με κάποια νέα τμήματα και πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η βασικότερη πηγή μετρήσιμων σφαλμάτων είναι η εκταμείευση μη επιλέξιμων δαπανών, έργων ή ε, συμμετεχόντων και δικαιούχων. Μιλάμε για ένα 65% όλων των μετρήσιμων σφαλμάτων και 74% του συνολικού ποστού λάθος. Παραδείγματο χάρη έχουμε μη επιλέξιμους συμμετέχοντες, υπερβολική χρέωση δαπανών προσωπικού ή ε, λανθασμένος υπολογισμός λειτουργικού κόστους. περισσότερες, περισσότεροι από αυτούς τους κανόνες τόσοι άλλους έχουν καθοριστεί από τα ίδια τα κράτη-μέλη και είναι σε ορισμένες περιπτώσεις ε, περίπλοκη χωρίς να υπάρχει λόγος ή ακόμα και πιο αυστηρή από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, αυτό το οποίο αποκαλεί επιχρήσωμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο δεύτερο βασικός, ε, η δεύτερη βασική πηγή είναι η μη συμμόρφωση με τους κανόνες δημοσίων προμηθειών. Ε, αυτά αποτελούν γύρω στο 30% των μετρήσιμων σφαλμάτων και γύρω στο 25% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Σε αντίθεση με την ε, περιφερειακή πολιτική, όλα τα συμβόλαια τα οποία ελέγχθηκαν ήταν κάτω από το κατόφλι που ορίζουν οι οδηγίες. Εν ολίγης δηλαδή και πάλι εθνικοί νόμοι παραβιάστηκαν. Και για ζητήματα δημοσίων προμηθειών και επιλεξιμότητας παρατηρήσαμε πως οι ε, πως η επανάληψη των πληρωμών σε προβληματικά επιχειρησιακά προγράμματα σημαίνει υψηλότερο κίνδυνο. Επίσης βρήκαμε μετρήσιμα λάθη σε 5 από τις 8 συναλλαγές που ελέγχθησαν για ένα πρόγραμμα το οποίο είχε κλείσει χωρίς καμία δημοσιονομική διόρθωση κάτι το οποίο επιβεβαιώνει τα περσινά συμπεράσματά μας πως τα μη αξιόπιστα έγγραφα κλεισίματος μπορεί να οδηγήσουν σε μη τακτικές ε, καταβολές εξόδων εκτός αν η Κομισιόν λάβει διορθωτικές δράσεις σε επόμενη φάση. Το κεφάλαιο 6 συμπεριέλαμβανε το 2012 ένα νέο τμήμα για την χρήση των ε, απλοποιημένων επιλογών κόστους. Το συνέδριο πέρσι συνέστησε μεγαλύτερη χρήση των καταποκοπήν ε, ποσών αντί για την επιστροφή των όντως καταβληθέντων εξόδων. βασικός λόγος ήταν πως έτσι θα υπήρχε μικρότερο ποσοστό σφάλματος και θα μειώνονταν κατά πολύ και το διοικητικό βάρος. Από το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει διευρύνει τη χρήση τέτοιων πληρωμών. Ένα τέταρτο των συναλλαγών που ελέγξαμε δειγματοληπτικά το 2012 είχαν δηλωθεί με βάση αυτές τις απλοποιημένες επιλογές. Συναλλαγές αυτές αφορούν περίπου τα μισά από τα προγράμματα τα επιχειρησιακά που ελέγξαμε. Σημειώνουμε πως το συνέδριο δεν βρήκε μετρήσιμες ή μη, μετρήσιμα ή μη σφάλματα που αφορούν την συγκεκριμένη χρήση με καταποκοπήν ποσά. Φαίνεται έτσι πως επιβεβαιώνεται πως οι επιλογές αυτές προσφέρονται λιγότερο για λάθη, για σφάλματα και η πιο εκτεταμένη χρήση τους θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα στο ποσοστό σφάλματος. Κυρίες και κύριοι, παρά το ότι το κεφάλαιο 6 δεν περιέχει τμήμα για δημοσιονομικές διορθώσεις, οι δημοσιονομικές διορθώσεις είναι στο κεφάλαιο 1, όπου νομίζω πως η κύρια συζήτηση και θα το συζητήσουμε αύριο με τον εισηγητή. Θα ήθελα να εξηγήσω πώς λάβαμε υπόψη τις δημοσιονομικές διορθώσεις το 2012. Και αυτό θέλω να το κάνω γιατί είναι μεγάλη η έκταση και οι συνέπειε των διορθώσεων που επέβαλε η Γενική Διεύθυνση, ειδικά στη Ρουμανία. Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ συνεδρίου και κομισιών. Ε, καθώς προσεγγίζουμε το ζήτημα από διαφορετικές, αλλά θα έλεγα παραπληρωματικές ε, πρόπτικες. Το συνέδριο αξιολογεί την ομότητα και τακτικότητα κανονικότητα των δαπανών, ενώ το Κομισιόν είναι υποχρεωμένο να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της κοινότητας και βεβαίως οι διορθώσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο γι' αυτό. Πρέπει βεβαίως να σημειώσουμε πως λαμβάνουμε υπόψη τις δημοσιονομικές διορθώσεις, κάποιες από αυτές, όταν υπολογίζουμε το ποσοστό σφάλματος. Οπότε όταν βρίσκουμε ένα σφάλμα και έχει επιβληθεί εντός του ιδίου έτους δημοσιονομική διόρθωση σε επίπεδο έργου δεν συνυπολογίζεται αυτό στο ποσοστό σφάλματος. Όμως, οι καταποκοπήν διορθώσεις που δεν αφαιρούν από την δήλωση τις μη κανονικές δαπάνες στο επίπεδο έργου δεν επηρεάζουν το ε, ποσοστό σφάλματος που υπολογίζουμε. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον ε, καταποκοπήν 25% διόρθωση που επιβλήθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της Ρουμανίας όπως περιγράφεται στις στήλες 1 και 2 και παραγράφους 1.31 και 33 του κεφαλαίου 1 της ετήσιας έκθεσης. Τέλος, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων, Εστιαστήκαμε όπως και τα προηγούμενα χρόνια στον ρόλο που παίζουν οι ελεκτικές αρχές στα κράτη-μέλη και στη δουλειά που κάνει η Κομισιόν για να τα υποπτεύσει. Το τμήμα αυτό της εργασίας παρουσιάζεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 5 και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για την περιφερειακή πολιτική. Πρώτον, για τις ελεγκτικές αρχές το 2012 αξιολογήσαμε 4 από τις 112 αρχές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Συνεχίσαμε έτσι τη δουλειά που έχει ξεκινήσει από το 2010. Συνολικά 19 ελεγκτικές αρχές για το ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΚΤ ελέγχθηκαν σε 15 κράτη-μέλη. Το 2012 καταλήξαμε πως μία στις τέσσερις ήταν αποτελεσματικές και οι υπόλοιπες ήταν εν μέρη αποτελεσματικές. Στη δεύτερη περίπτωση βρήκαμε συγκεκριμένα προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο είχε διεξαχθεί ο έλεγχος ε, και αναφέρθηκαν τα αποτελέσματα της Κομισιόν Δεύτερον. Το συνέδριο βρήκε και κάποιους τομείς βελτίωσης όσον αφορά την εποπτεία των αρχών αυτών από την Κομισιόν. Τα προβλήματα αυτά τα βρήκαμε κυρίως ε, λόγω του ότι δεν υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες ε, στην Κομισιόν για να διεξαγάγει αποτελεσματικά τους ε, ελέγχους και τις εκθέσεις επί των εκθέσεων των ελεκτικών αρχών. Επίσης δημοσιεύσαμε το Δεκέμβριο στην σελίδα μας την ειδική εκθέση 16-2003 που λέγεται «Απολογισμός του ενιαίου ελέγχου και το πώς η Κομισιόν βασίζεται στις εθνικές αρχές στον τομέα της συνοχής». Η έκθεση αυτή κάνει αυτό το οποίο λέει ο τίτλος της. Σύμφωνα με το άρθρο 73 του κανονισμού 1083. Ε, και κάλυπτε την περίοδο 2010 μέχρι τέλος 2012. Συνοψίζοντας, πρέπει να σημειώσουμε πως ο βαθμός και οι συνέπειες των προβλημάτων που περιγράφονται και στο κεφάλαιο 5 και στην ειδική έκθεση υπαριθμών 16 του 2013 ήταν, είχαν μικρότερη κλίμακα στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, the member of... Να ευχαριστήσουμε πολύ το μέλος από το Λεκτικό Συνέδριο, τον κύριο Λάζαρο Λαζάρου. Σας ευχαριστούμε για τη δήλωσή σας αυτή. Ευχαριστώ να δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Επίτροπο για να κάνει την εισαγωγή του. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω λέγοντας καταρχάς ότι εκτιμώ πάρα πολύ την επικοδομητική σχέση που έχουμε με το Ελεκτικό Συνέδριο, καθώς επίσης και την ισορροπημένη αυτή έκθεση από το Ελεκτικό Συνέδριο που έχουμε μπροστά μας σήμερα. Μέσω της έκθεσης αυτής βλέπουμε πραγματικά ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος και βλέπουμε ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι περήφανος που ο τομέας της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων είναι ένας τομέα ο παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό σφάλματος. Μπορεί να βρισκόμαστε πάνω από το 2%, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι το ποσοστό σφάλματος δεν αντικατοπτρίζει την κατακοποπή, με συγχωρείτε, διόρθωση που έχουμε για το 2012 για τη Ρουμανία, 25%. Ο προπολογισμό αυτό, μόλον ότι μπορεί να μην διορθώνει ακριβώ τα ποσά τα οποία υπάρχουν σε κάθε σχέδιο, είναι αποτελεσματικό από οικονομική πλευρά. Και βλέπουμε ότι για τρίτη συνεχόμενη φορά ανταποκρινόμαστε στους στόχους που έχει θέσει η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε πραγματικά να επαληθεύουμε και να κάνουμε τους κατάλληλους ελέγχους. Ποιες είναι οι βασικές συστάσεις που κάνει το συνέδριο. Στην έκθεση του 2012 βλέπουμε ένα ξεκάθρο μήνυμα όσον αφορά την απλούστευση. Εν 26 περίπου της 100 των προγραμμάτων του ESF που έχουν ελεγχθεί από το συνέδριο αποτελούν και χρησιμοποιούν μία περισσότερες μορφές απλούστευσης, ενώ το συνέδριο δεν έχει εντοπίσει κανένα σφάλμα όσον αφορά τα προγράμματα αυτά τα οποία χρησιμοποιούν τις απλουστευμένες μορφές κόστους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η απλούστευση την οποία έχουμε προωθήσει πάρα πολύ αποτελεσματικά πέρα από το ότι μειώνει την, το γραφειοκρατικό άχθος, και κάνει τελικά τα προγράμματα πιο αποτελεσματικά, μειώνει επίση και το επίπεδο σφάλματο. Για το ζήτημα λοιπόν αυτό και όσον αφορά και το gold plating, τον κανονιστικό υπερθεματισμό, μπορούμε να πούμε ότι η Γενική Διεύθυνση Απασχόληση έχει υποβάλει και μια σύντομη έκθεση προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί θα δείτε συγκεκριμένα παραδείγματα και δράσει που έχουν αληφθεί από κοινού με τα κράτη-μέλη, προκειμένου πραγματικά να επιφέρουμε θετικά αποτελέσματα και να τροποποιήσουμε αποτελεσματικά τα πράγματα. Συμφωνούμε με το συνέδριο ότι θα πρέπει βάσει τη εμπειρία αυτή να συνεχίσουμε. Να υπάρχει μια ανταλλαγή των πρακτικών και ο νέο κανονισμό που έχει υιοθετηθεί μα δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να προωθούμε ενεργά τι συστάσει του ελεγκτικού συνεδρίου για να φτάσουμε περίπου στο 50% των προγραμμάτων ESF που θα χρησιμοποιούν το σύστημα SEO, δηλαδή επιλογές απλουστευμένου κόστους μέχρι το 2018 συγκεκριμένα. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην επαλήθευση των ελέγχων. Για το ζήτημα αυτό έχει υποβληθεί σχετική έκθεση από τη Γενική μου Διεύθυνση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία εξηγείται ποιε ακριβώ είναι οι δυναμίε που έχουμε εντοπίσει και πώ εμεί θα τι αντιμετωπίσουμε ζητούμε από τα κράτη-μέλη να πετύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στον τομέα αυτό. Σίγουρα μπορούν να γίνουν περαιτέρω διορθώσει στη νέα περίοδο προγραμματισμού, τη νέα δημοσιονομική περίοδο. Πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι ακόμα πιο αποτελεσματικοί και πιο αυστηροί στο πρωτογενέ, στο πρώτο επίπεδο ελέγχου. Τέλο, θα ήθελα να αναφερθώ και στο έργο που επιτελούν οι ελεγκτικές αρχέ. Θα συνεχίσουμε με μια προσέγγιση που θα βασίζεται στο κίνδυνο και θα επικεντρωθούμε κυρίως σε αυτές τις ελεγκτικές αρχές οι οποίες παρουσιάζουν ένα υψηλό προφίλ κινδύνου. Ως προς αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για την έκθεση την οποία επέβαλε το 2013 όπου αναλύει περισσότερο τις εκθέσεις ελέγχου που έχουν υποβάλει τα κράτη-μέλη. Βλέπουμε επίσης πώς μπορούμε να εντάξουμε περισσότερο στην έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε εκθέσεις που υποβάλλουν οι εθνικές ελεγκτικές αρχές. Πιστεύω ότι το πόρισμα της έκθεσης αυτής θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια σφαιρική αποτίμηση των ελεγκτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, όσον αφορά την ορθή χρήση των πόρων του ESF, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια πάρα πολύ αυστηρή πολιτική όσον αφορά την διακοπή πόρων. Ένα 38 συγκεκριμένα πληρωμές κατά το παρελθόν έτος προς δύο κράτη-μέλη αναστάλθηκαν. Το 2013 ήταν 29 τα προγράμματα αυτά τα οποία σταμάτησαν ενώ έπρεπε να αναστείλουμε 11 προγράμματα, να στείλουμε την πληρωμή για 11 προγράμματα. Τα κάνουμε όλα αυτά προκειμένου να προστατεύσουμε τον κοινοτικό προπολογισμό. Μεταξύ του Ιανουαρίου και του Δεκεμβρίου του 2011 η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης χρησιμοποίησε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ ως ποσό διορθώσεων για όλα τα προγράμματα ενώ το 2012 το ποσό αυτό ήταν 400 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πολύ αυτή αυστηρή πολιτική δεν έχει εμποδίσει σε καμία περίπτωση την απορρόφηση. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τα δύο τρίτα του συνολικού ποσού για την περίοδο 2007-2013 ήδη είχαν ε, δαπανηθεί μέχρι τα τέλη του 2013 και αν πάρουμε μόνο το έτος 2013 βλέπουμε ότι 13,8 δισεκατομμύρια ευρώ είχαν ε, δαπανηθεί με μια αύξηση 22% σε σχέση με το παρελθόν έτος το 2010. Κυρίες και κύριοι, δεν έρχομαι εδώ πέρα σήμερα για να σας πω ότι τα πάντα είναι τέλεια. Η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου καταδεικνύει ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν, να αντιμετωπιστούν. Βλέπουμε ξεκάθαρα όμως ότι έχει επιτευχθεί μια σημαντικότατη πρόοδος προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε την κανονικότητα και ορθότητα των δαπανών μας. Μπορούμε λοιπόν να βασιστούμε στην πρόοδο αυτή που έχει επιτευχθεί, προκειμένου να έχουμε πιο αποτελεσματικές και πιο ποιοτικέ επαληθεύσεις για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, εκατομμύρια ανθρώπων που είναι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίοι απαιτούν από εμά να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε ευρώ από τον κοινωνικό προπολογισμό προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο από μόνο του δεν μπορεί να επιλύσει το ζήτημα τη υψηλή ανεργία, ούτε καν τη ανεργία των νέων γιατί υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι που οδηγούν στην ενεργία αυτή. Πάντως το ESF μπορεί να συμβάλλει πολύ σημαντικά. Από το 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει βοηθήσει 68 εκατομμύρια Ευρωπαίους και θεωρούμε ότι η υποστήριξη αυτή από το ESF έχει οδηγήσει σε 5,5 ε, νέες θέσεις εργασίας, 5,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας υπάρχουν 5,5 εκατομμύρια άτομα τα οποία κατάφεραν μέσω των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ESF βοηθά ενεργά τους ε, Ευρωπαίους πολίτες να καταφέρουν να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα εποχή τεχνολογικών αλλαγών και να αντιμετωπίσουν επίσης την ε, σφοδρότατη αυτή οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, λέει Πρόεδρος, στα γερμανικά τώρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα δώσω τώρα τον λόγο στον εισηγητή μας. Τον λόγο έχει λοιπόν ο κύριος Μάρκος Πίπερ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αγαπητό μέλος του Ελληνικού Συνεδρίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Η νομότητα των δαπανών, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Επίτροπος, δεν είναι νομίζω ζήτημα επίμαχο και δεν αναμπαίνονται βεβαίως εκεί διαμάχες, αλλά όσον αφορά την μέθοδο βεβαίως είναι ανοιχτό το ζήτημα του γιατί το ποσοστό του σφάλματος ε, που διαπιστώθηκε στο 2,2 ανέβηκε στο 3,2%. Ποιες είναι οι αιτίε γι' αυτό. Η Κομισιόν πιστεύει πως ε, θα, είχε, θα έπρεπε να έχει μείνει το ίδιο, αλλά Βεβαίως ο καθένας εδώ πέρα έχει τα επιχειρηματά του. Αυτό το οποίο θα θέλαμε εμείς για το μέλλον είναι να υπάρξει μια κοινή τοποθέτηση Κομισιών και Ελεγκτικού Συνεδρίου έτσι ώστε να έχουμε και μεθοδολογικά κάποια περαιτέρω βοήθεια για να μπορέσουμε να κρίνουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πλαίσιο αυτό Εδώ πέρα το συνέδριο λέει πως μία σύσταση από το έτος 2009-2010, μία μόλις υιοθετήθηκε πλήρως από την Κομισιόν. Πέντε ακόμα υιοθετήθηκαν μερικώς, ε, άλλη μία επίσης, ε, ο λίγον τι και οι υπόλοιπες καθόλου. Οπότε θα ήθελα το ελεγκτικό συνεδρίο να μας πει τι αναμένει συγκεκριμένα επ' αυτού και ίσως μετά η Κομισιόν να μας δώσει μια απάντηση στην κριτική του συνεδρίου. Όπως είπαμε όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν εδώ και κάποια χρόνια και οπωσδήποτε ε, κάποια απάντηση περιμένουμε. Κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο με ανησυχεί όμως πολύ περισσότερο είναι... δεν είναι τόσο το ποσοστό του σφάλματος αλλά το ποσό του φάλματος βασίζεται σε τελική ανάλυση στα στοιχεία που δίνουν τα κράτη-μέλη και σύμφωνα με την άποψη του ελεγκτικού συνεδρίου η εμπιστοσύνη που μπορούμε να δείξουμε σε αυτά είναι περιορισμένη και αναφέρομαι εδώ πέρα σε έκθεση της ίδιας της Κομισιόν, λεγόμενη Γενική Επισκόπηση των Αποτελεσμάτων Θεματικού Ελέγχου ε, σύμφωνα με για επί των ελέγχων που έκαναν τα κράτη-μέλη εκεί πέρα. Αναφέρεται πως οι ελεγκτικές αρχές έχουν σοβαρές ελλείψεις, η οργάνωση και η επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικών αρχών και ελεγχομένων είναι προβληματική. Συνεχώς οι ίδιες παραβιάσεις όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες δεν υπάρχει διοικητική ικανότητα κλπ. λοιπά. Αυτά που σας διαβάζω είναι από έκθεση της ίδιας της Κομισιόν, έτσι. Οπότε, ανησυχώ κάπως, εξού και το ερώτημά μου προς τον κύριο Επίτροπο. Εντάξει, ποστό σφάλματος 2,2%. Καλώς, αλλά πόσο αξιόπιστο είναι αυτό το οποίο σας στέλνουν τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το πρώτο. Μια δεύτερη ερώτηση για αυτή την κανονιστική υπερβολή. Εδώ πέρα υπάρχουν διαφορές σοβαρές μεταξύ των κρατών μελών. Βλέπουμε πως η Κομισιόν έχει αρκετά μεγάλη εξουσία εδώ πέρα και θα μπορούσαν να αποφευχθούν κάποια απλά λάθη, αλλά πού ε, οφείλονται αυτές οι μεγάλες ε, διαφορές. Έχει κάποια ιδέα η Κομισιόν. Μετά, ένα ερώτημα όσον αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων. Εντάξει, ε, ομολογώ ότι είναι άδικο, δεν ήταν αυτός γραπτές ερωτήσεις, αλλά είναι μια καθημερινή πολιτική συζήτηση που την κάνουμε. Δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχουμε ένα ποσοστό μεταξύ 30 ή 50 ή όταν είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα 60% ποσοστό απορρόφησης. Αυτά γράφονται στις εφημερίδες. Δηλαδή υπάρχουν δισεκατομμύρια ευρώ που παραμένουν αχρησιμοποίητα. Ποια είναι η αιτία κατά την άποψη της Κομισιόν. Ειδικά αν δούμε το τι γίνεται στη Ρουμανία ή στη Βουλγαρία αλλά και στη Γερμανία όπου σε μεγάλες πόλεις έχουμε τεράστια προβλήματα. Αν υπάρχουν τα λεφτά γιατί δεν ε, χρησιμοποιούνται. Ποια είναι η αιτία. Και τελευταία παρατήρηση Θα ήθελα να αφαιρθώ και πάλι στο ότι όσον αφορά την ε, νομιμότητα των ε, δαπανών, τουλάχιστον τυπικά, ε, τα πάντα είναι εντάξει, αλλά κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για το ότι βοηθήσατε στην διατήρηση 5,5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας και 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τώρα περισσότερα προσόντα. Να το δούμε πανευρωπαϊκά. Όπου μιλάμε σε κάποια κράτη-μέλη για ανεργία των νέων πάνω από 50% και ανεργία μεταξύ 20 και 30% γενική. Και ταυτόχρονα λάβουμε υπόψη πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αυτή τη λεγόμενη ε, εγγύηση για την νεολαία. Α, ρωτιέμαι. Αν τα λεφτά αυτά πραγματικά χρησιμοποιήθηκαν αποτελεσματικά ώστε να μπορέσουμε να πούμε πως εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε και μπορούμε να δώσουμε μια εγγύηση τώρα στην νεολαία. Εγγύηση στην νεολαία σημαίνει πως ε, ο καθένας μέχρι μια κάποια ηλικία θα έχει μια θέση είτε απασχόλησης, είτε εκπαίδευσης, είτε κατάρτισης. Αυτό εγγυάται η Ευρώπη. Εσείς στην απάντησή σας κάπως πήρατε πίσω αυτή την υπόσχεση. Πλέον δεν μιλάτε για εγγυήση, αλλά για μια υπόσχεση. Υπόσχεση να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας οι άνεργοι νέοι. Ε, μια υποχώρηση από πλευρά σας πριν λέγατε πως δίνουμε εγγύηση. Εγώ θεωρώ πως το πρόγραμμα αυτό πρέπει να έχει ένα ακόμη πιο ειλικρινές όνομα. Γιατί, Γιατί δημιουργούμε προσδοκίες ε, που ποτέ δεν θα μπορέσουμε να τηρήσουμε. Και δεν απαντήσατε λοιπόν στο ερώτημα ποιο είναι το ποσοστό των κονδυλίων του κοινωνικού ταμείου που χρησιμοποιήθηκαν για μέτρα εκπαίδευσης, ε, διατήρησης της απασχόλησης, ποιο ποσοστό από αυτά πήγε σε αυτά τα κεφάλαια. Δεν ξέρω. Ε, αν είναι 70-80% θα μου πείτε. Και μετά το ερώτημα είναι κατά πόσο μειώσαμε την ανεργία των νέων και την ανεργία συνολικά. Προφανώς ανέβηκε η ανεργία και ειδικά η ανεργία των νέων. Οπότε πρέπει να πω πως δυστυχώς η διακηρύξεις σας ε, νομίζω αντιφάσκουν με το αποτέλεσμα. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν μιλάμε για εγγυήσει από πλευρά Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στο μέλλον. Τελευταία παρατήρηση αφορά πάρα πολλές δραστηριότητες, ε, όπως παραδείγματος χάρη οι συστάσεις αναχώρα, όπου μπαίνετε στην εθνική νομοθεσία και λέτε πως ε, τα συνταξιδοτικά συστήματα δεν είναι σωστά ή ασκείτε κριτική στα επιδόματα παιδιών και άλλα τέτοια. Οπότε αναρωτιέμαι πραγματικά λαμβάνετε υπόψη την αρχή του κοινωνικού κράτους η οποία υπάρχει στα περισσότερα συντάγματα των κρατών μελών. Πώς μπορούμε, ως, πώς μπορείτε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπαίνετε σε αυτά τα χωράφια. Έχω, δεν μπορώ να αξιολογήσω το εάν οι δυνατότητες που έχει η υπηρεσία σας πραγματικά ανταποκρίνονται στην εντολή σας ή εάν με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνετε εθελοντικά σπαταλάτε πόρους οι οποίοι θα ήταν καλύτερο να διατεθούν για τον έλεγχο των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παραδείγματο χάρη να ανεβούει ο αριθμός των διπλωματών δειγματοληπτικών ελέγχων και να μην βασίζεται μόνο στα κράτη-μέλη. Εγώ λοιπόν θα ήθελα ισχυρότερη Ευρώπη και μια κομισιόν η οποία δεν θα την κάνουν ό,τι θέλουν τα κράτη-μέλη αλλά ειδικά στα θέματα ελέγχου και υπεύθυνη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων, θα ασχοληθεί με τις ελλείψεις που αναφέρετε οι ίδιοι κύριε Επίτροπε στην έκθεσή σας και θα ασχοληθείτε πολύ περισσότερο. Οπότε, επαναλαμβάνω, ε, η μομφή λοιπόν δεν αφορά την ε, νομότητα των δαπανών αλλά στο ότι βασιζόμαστε πάρα πολύ στα κράτη-μέλη και εδώ πέρα νομίζω συμφωνούμε με τους περισσότερους συναδέλφους ε, πως θέλουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή απάντηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και Σιγητά. Θα δώσω τώρα τον λόγο στα μέλη της Επιτροπής και στους συντονιστές. Η κυρία Γκρέσλε πρώτη. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Πάντα χαιρόμαστε ε, όταν έρχεστε. γιατί είστε αρμόδιος για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, τις κοινωνικές δαπάνες στο κοινωνικό ταμείο. Ήδη πέρσι είχαμε έντονες συζητήσεις για το τι γίνεται με τα λεφτά για την ανεργία των νέων. Τώρα εντωμεταξύ εγώ ρώτησα πάρα πολλές ε, ΜΚΟ που έλαβαν λεφτά και μου είπαν πως δεν ε, ήξεραν γιατί δεν κρατάει κανείς ε, στοιχεία. Οι δε ίδιες οι ΜΚΟ μου λένε «Μα εμείς όλη μέρα στοιχεία κρατάμε και τα στέλνουμε». Κοιτάξτε, οι ίδιοι, οι ίδιοι δικαιούχοι λένε πώς θα στέλνουν τα στοιχεία. Για μένα το ερώτημα είναι απλό. Πού είναι αυτά τα στοιχεία. Για μένα είναι σημαντικό το θέμα για να μπορέσουμε να πούμε ότι είχαμε και μια επιτυχία. Το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, μια ομάδα την οποία είχαμε προβλήματα στη Γερμανία που είναι η Ρωμά. Και το ζήτημα ακριβώς είναι η ροή κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προς τη μειονότητα αυτή και βλέπουμε μετά πως σε Βουλγαρία και Ρουμανία είναι πολύ χαμηλή η ροή. Δηλαδή είναι τόσα χρόνια κράτη-μέλη αυτές οι χώρες. Και βλέπουμε πως τα κονδύλια για Βουλγαρία και Ρουμανία είναι, η εκταμίευσή τους είναι κάτω από 10%. Ποια είναι η αιτία και τι κάνει η Κομισιόν για να αυξηθεί η απορρόφηση των ε, κονδυλίων. Είδα τα νούμερα και σας ευχαριστώ. Τι γίνεται αυτή την στιγμή. Βεβαίω μιλάμε για Βουλγαρία για μια αύξηση 57% και στη Ρουμανία 41%. Αλλά αυτό είναι προκαταβολές, έτσι. Το ζήτημα είναι επίσης τι επιτυγχάνουμε, τι έχουμε καταφέρει με τους Ρωμά, με την ένταξή τους. Πρέπει να απαντήσουμε στους ψηφοφόρους μας έτσι, γιατί αυτό είναι και το νόημα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Να γίνεται κάτι με αυτά τα λεφτά. Αυτό ανησυχώ πάρα πολύ. Για το ότι δεν μπορεί να μας πει τίποτα η Κομισιόν για το θέμα. Οπότε πραγματικά σας παρακαλώ να το δείτε χρειαζόμαστε αυτές τις ε, πληροφορίες. Δεν ερχόμαστε εδώ πέρα για να πούμε μετά στους ψηφοφόρους μας ούτε και εγώ ξέρω. Μετά, ένα τεχνικό αλλά και πολιτικό ταυτόχρονα ερώτημα όσον αφορά τις προκαταβολές αυτές. Από πότε είναι ακριβώς αυτά τα ποσά και ποιο είναι το ύψος, ε, το ύψος τους. Διαπιστώσαμε πως πάνω από το 25% των, ε, των 20% με των προκαταβολών ε, της Κομισιόν είναι πάνω από 6 χρόνια πριν. Αυτό δεν αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο βεβαίω μόνο. Επίσης, να σας πω, υπάρχει και μια στρατηγική για τους Ρωμά. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή τη στρατηγική, εάν πουθενά εδώ πέρα δεν μας έχετε υποβάλει τίποτα. Ποια είναι τα αποτελέσματα κατά την άποψή σας όσον αφορά την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τι προγραμματίζει η Κομισιόν όσον αφορά μια αξιολόγηση ex των εθνικών στρατηγικών ε, πλαισίου και των εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τι προγραμματίζεται για να επιτύχουμε κάτι για αυτή την ομάδα ανθρώπων. Δεν μπορούμε να πούμε στους ψηφοφόρους μας ε, πως ε, πληρώνει ο ευρωπαϊκός προπολογισμό και ξαναπληρώνουμε μετά στη Γερμανία για την ένταξή τους γιατί προφανώς δεν είμαστε σε θέση να βασιστούμε στα κράτη-μέλη είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και ξέρετε ε, είναι λυπηρό το ότι πράγματι υπάρχει αυτή η παρεξήγηση όσον αφορά την ε, ελεύθερη διακίνηση και στον ε, γερμανικό τύπο αλλά είναι κάτι βεβαίως το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους Γερμανούς ψηφοφόρους. Σας ευχαριστώ, Γιάννης Γκάια. κάτι παρόμοιο κι εγώ με αυτό το οποίο είπε η κυρία Γκρέσλε έχω να πω αλλά το ερώτημα μου προς τον Επίτροπο αφορά την ε, σχέση Διακοπή της ε, χρηματοδότησης και επίτευξη των στόχων. Πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η προτεραιότητα του Κοινοβουλίου στα κράτη-μέλη. Μέχρι τώρα η προτεραιότητα τη Επιτροπής μας ήταν η νομότητα των δαπανών. Σε κάθε διαδικασία απαλλαγής ε, ε, την οποία έχω παρακολουθήσει ζητούσαμε από την Κομισιόν να διακόψει τα προγράμματα εάν δεν ήταν εγγυημένη νομιμότητα των δαπανών. Εάν το κάνει όμως αυτό η Κομισιόν, κάτι το οποίο μέχρι τώρα βεβαίως χειροκροτούσαμε και δεν πάνε τα λεφτά εκεί όπου θα έπρεπε γιατί βεβαίως ε, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την νομιμότητα των δαπανών, ο πολιτικός στόχος δεν επιτυγχάνεται. Η υποψία μου είναι πως η λύση του ενίγματος είναι αυτό το οποίο ανέφερε η συνάδελφος με τις ε, χώρες που ανέφερε, Βουλγαρία και Ρωμανία. Πρέπει λοιπόν να κρίνουμε τι είναι σημαντικότερο να έχουμε νομότα των δαπανών και να μην πάνε τα λεφτά. Αλλά τότε δεν θα επιτευχθεί ο πολιτικός στόχος ένταξη των Ρωμά. Ή ε, είναι ο πολιτικός στόχος, ο σημαντικός στόχος. Κοιτάξτε, δεν, λέω ότι το ένα αποκλείει το άλλο. Μα αυτό συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να σκεφτούμε αν είναι αυτή η μομφή, όπως το είπες, προς την Κομισιόν, έχουμε ένα δίλημα, γιατί υπάρχει ο πολιτικός στόχος και οπότε θα πρέπει να δεχτούμε το υψηλότερο ποσοστό σφάλματος ή αλλιώς θα πέσει το ποσοστό σφάλματος και κακοδιοχείρισης για να επιτύχουμε το στόχο. Ε, αλλιώς, ε, εντάξει κάτι πάντα θα βρούμε για να βρίζουμε την Κομισιόν, αλλά δεν είναι και πολύ δίκαιο, έτσι για να το πω λίγο χοντρά. Ε, κοίτα, ε, ε, τώρα μην φτιάχνει διαφωνίες από εκεί που δεν υπάρχουν. Εγώ θέλω να προτείνω λύση. Είχα συζητήσει και με έναν ε, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βάδης Βιρτεμβέργης, τον οποίο τον πέτυχα στο Βουκουρέστι γιατί θα έστελνε υπαλλήλου του για να βοηθήσουν τη διοίκηση. Ε, εκεί πέρα νομίζω είναι η λύση. Και εδώ πέρα θα με ενδιέφερε η άποψη του κυρίου Άντορ. Πώς το βλέπει, πώς βλέπει δηλαδή τη σχέση ε, επίτευξης ε, πολιτικών στόχων και νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών. Εάν έχουμε βρεθεί στη δύσκολη θέση που περιέγραψα, θέλω να μάθω τι σκέφτεται η Κομισιόν για να βγούμε από αυτήν. Σας ευχαριστώ. Να ρωτιέμαι Μήπω το ότι η ένταση αυτή οφείλεται στο ότι είμαστε στο 2014 και όχι στο 2012. Τέλος Ο κύριο Μούλτερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μπαίνει κανεί σε πειρασμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται όσον αφορά την αγορά εργασία και τους ε, Βούλγαρου και τους Ρουμάνους ε, αλλά εγώ θα αντισταθώ σε αυτόν τον πειρασμό. Δεν είναι τώρα η ώρα γι' αυτό. κάποιε άλλε ερωτήσει, ερωτήσεις γενικότερο χαρακτήρα πρώτα-πρώτα. Σε σχέση με την ε, κοινωνική πρόνοια, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πιο αξιοθαύμαστα συστήματα είναι η εφαρμογή των ε, ε, δημοσιονομικών διορθώσεων που τα καταφέρατε πέρσι να μειώσετε το βαθμό σφάλματος εντυπωσιακά. Βέβαια ξέρουμε πώς κάνει τον υπολογισμό του το ελεκτρικό συνέδριο και αν είχε το 25% της Ρουμανίας βάλει μέσα τότε θα είμαστε στα ίδια επίπεδα. Αυτό είναι ένα παράπονο το οποίο το έχω ακούσει από όλους σε όλες τις ε, συζητήσεις με τους ε, επιτρόπους. Για πετε μας, σκοπεύετε να κάνετε κάτι κατά του ελεκτρικού συνεδρίου γιατί το θέμα είναι ότι το Ελληνικό Συνέδριο τηρεί τι διεθνεί προδιαγραφέ, του διεθνού κανόνε. Οπότε η ερώτησή μου είναι, ποια είναι τα επιχειρήματα τόσο ώστε να παρεκκλίνει κανείς από αυτούς τους διεθνείς κανόνες, τους οποίους και επικαλείται και χρησιμοποιεί το ίδιο Συνέδριο. Δεύτερη ερώτηση τώρα είναι η εξή. 2% είναι αυτό το μαγικό όριο. Αν κανείς είναι κάτω από το 2% τότε είναι άψογος. Αλλά για πέστε μας. Τι μας εμπόδιζε, τι σας εμπόδιζε να μην μπορούμε να κατέβουμε κάτω από το 2% όσον αφορά το επίπεδο σφάλματος. Κύριε Γκρέσλε, επόμενο. Θέλω μόνο να ξεκαθαρίσω πως δεν βοηθάει τους Ρωμά να πάρει ένα ΜΚΟ τα λεφτά που δεν έχει σχέση με το αντικείμενο ή κάποιος άλλος ο οποίο δεν έχει σχέση με το αντικείμενο. Μα όταν έχουμε απάτη ή οτιδήποτε άλλο οδηγεί την Κομισιόν στο να παγώσει τα κονδύλια όπως έγινε σε πέντε ρουμανικά προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων το 2012 δεν, δεν βοηθάει τίποτα. Έτσι. Ε, η δουλειά μας εδώ πέρα, και εγώ δεν το έχω ποτέ πει έτσι, δεν είναι να ψάχνουμε πράγματα για να ασκούμε κριτική στην Κομισιόν και ποτέ δεν το έκανα αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι, και γι' αυτό ακριβώς ρώτησα, γιατί είναι τόσο περιορισμένη η ε, ροή. Αυτό. Αλλιώς θα ήμουν και εγώ πολύ ευχαριστημένη. Ευχαριστώ κύριε Αντρέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλούμε τώρα για αυτή τη διόρθωση, το κατά πόσο έχει δεν έχει επιπτώσεις όσον αφορά το επίπεδο σφάλματος. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, θεωρώ ότι αυτή η διόρθωση μόνο καλό μπορεί να κάνει σε αυτό το επίπεδο σφάλματος. Εφόσον επιστρέφονται κάποια χρήματα από τον τελικό δικαίου και όταν έχουμε αυτό το, το, το αυτό το καταποκοπήν ε, ποσό και έχουμε τη διόρθωση, τότε έρχονται τα χρήματα από την ε, σχετική κυβέρνηση, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουν ανακριθεί από τον ε, από τον, από τον επιλέξιμο, από τον δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος έχει πληρώσει δύο φορές. Άρα οι διορθώσεις έχουν ή δεν έχουν επιπτώσεις ε, επί του, επιπέδου φάρματος. Δεν έχουν, δεν έχουν προέλθει από τον ε, από τον τελικό ε, αποδεκτή δικαιούχο. Και οποίο για Ορμανία, Βουλγαρία θα, θα, θα, θα είχαν κάποια διαφορετικά αποτελέσματα επιτύχει εάν υπήρχε άμεσο έλεγχο όταν δεν παίρνουν τα ταμεία από το κοινωνικό ταμείο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο το οποίο ε, οφείλουν, στο οποίο πρέπει να υπάρχει για να μπορούμε να ασκήσουν σχετικού ελέγχου. Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο τον λόγο. Οπότε θα δώσω λόγο στον κύριο Επίτροπο για να απαντήσει όσο μπορεί. Έτσι, μπορείτε να μας στείλετε και άλλες απαντήσεις αργότερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω όσο μπορώ αγαπητοί κύριοι βουλευτές. Όσον αφορά τις ε, ερωτήσεις που έχετε θέσει, και πρώτα πρώτα, επιτρέψτε να σας πω πώς θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό να πιστώνουμε ότι υπάρχει ε, κάποια εκτίμηση θετική όσον αφορά αυτό το χαμηλό βαθμό σφάλματος, το οποίο δεν αφορά μόνο τη χρήση 2012, αλλά μια σειρά χρήσεων. Και κατά αυτές τις χρήσεις έχουμε τους υπολογισμούς της Διεθνής επασχόλησης αλλά έχουμε και τις εκτιμήσεις του Ελληνικού Συνεδρίου που κατατείνουν στο ίδιο αποτέλεσμα στην ίδια κατάληξη. όμω. θα πρέπει να δούμε τι θα, θα γίνει όσον αφορά τη συζητούμενη χρονιά, τη συζητούμενη χρήση του 2012. Όπω είπε το Ελληνικό Συνέδριο, ακόμη έχουμε θέμα, ακόμη έχουμε θέση να αμφιβόλω τη μεθοδολογία. Οπότε πρόκειται ουσιαστικά για κάτι το νέο, νέα εμπειρία και είναι κατανοητό ότι γίνεται μια τέτοια συζήτηση και θα πρέπει να δούμε τι καινούργιες διαστάσεις ξανοίγονται. Δεν καταλήξαμε ακόμα πουθενά, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορούμε παρά να έχουμε θεωρήσει θετικό το πόσο το συνέδριο έχει ταχθεί υπέρ της δικής μας μεθοδολογίας σε σχέση και με τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται από τις τραπέζης επίσης από τη συζήτηση κατεδείχθη σαφώς ότι για την ελόγω χρήση περίπου κατά το 40% του εφαρμόζου πρόκειται από μία και μόνο χώρα, τη Ρουμανία. Και βεβαίως προτίθεμαι να απαντήσω στις σχετικές ερωτήσεις, αλλά πρώτα πρώτα να σας τονίσω ότι παρά την εγκύτερη, την ιστορική, για την οικονομική. Κάθε χώρα είναι διαφορετική, πολλές φορές ε, δικαιολογείται να βάζουμε την Βουλγαρία και την Ρουμανία στο ίδιο καλάθι, ιδίως όσον αφορά το ότι μαζί μπήκαν αυτές οι δύο χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί προσεχώρησαν. Όμως, όσον αφορά το θέμα του υπέδου απορρόφησης, αλλά επίσης όσον αφορά και την ποιότητα της ε, απορρόφησης δεν βρίσκονται στην ίδια κατηγορία. Η Βουλγαρία προσφάτως έχει δείξει πιο καλό ρυθμό απορρόφησης. Άρα δεν υπάρχουν τα ίδια προβλήματα, δεν υπάρχουν κάποιες διακοπές, δεν υπάρχουν αναστολές, διακοπές στη χώρα αυτή. για την ανάκτηση επίσης ε, καυκίσματα μπροστά. Μιλάμε για 57,5% στη Βουλγαρία. Το οποίο δεν απέχει πολύ από το 66% του μέσου Ενώ η Ρωμανία είναι στο 41%. Επίση Επίσης, ε, για πάρα πολύ σημαντικό το ότι η πιο κοντινή χώρα σε αυτήν την κατάταξη, πιο κοντινή στην Ρουμανία, είναι το 48% που έχει η Σλοβακία. Πιο μακριά από λοιπόν αυτέ τι χώρε από το μέσο όρο. Επίση, σα σημαίνει επιζώτη. Καταρχήν τη σχετική περίοδο είχαμε την Ελλάδα, η οποία δεν τα πήγε τόσο καλά με το ρυθμό απορρόφηση ε, και είχε και βέβαια και τι ε, άλλε δυσκολίε. Όμω ε, αφιερώθηκε ενέργεια, αφιερώθηκε χρόνο από τη Γενική Διεύθυνση απασχόληση και έτσι να βελτιωθεί η απορρόφησε ε, και ποσοτικά και ποιοτικά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, τι δραστηριότητε ε, καλύπτουμε. Μιλούμε για εκτεταμένη συνεργασία όσον αφορά την κατάρτιση του προσωπικού, μιλούμε για δυνατότητε τη διοίκηση και για όλε αυτέ τι χώρε αλλά και για τη Ρουμανία το επίπεδο του σφάλματος αφορούσε την κατάσταση του προσωπικού, αναδιοργανώσεις κλπ. Στη Δερούμενη έγιναν κάποιες προσπαθίες ε, εδώ και ένα χρόνο περίπου, λίγο παραπάνω με την καινούργια κυβέρνηση, οπότε απεφασίστη να ε, εφαρμοστεί στην πράξη αναδιοργάνωση και εμείς ε, επιμείναμε κατά αυτή τη διαδικασία. Προσοχή να μην ε, έχουμε απώλειες όσον αφορά κάποιους ε, έμπειρους υπαλλήλους. Ενθάρρυνση, αλλά δεν σταυρώσαμε τα χέρια. Η Ρουμανική κυβέρνηση πήρε στα σοβαρά τις συμβουλές μας και τις προτάσεις μας, οπότε θα πρέπει να δούμε στο άμεσο μέλλον ποια είναι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία θα πετύχουν. Τώρα, για ποιες χώρες που αναφέραμε, πέραν της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, αλλά όσον αφορά την Βουλγαρία και για άλλες δύο χώρες, την Ουγγαρία, αλλά και την Τσεχία. Εν προκειμένου, η υλοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου για την εφαρμογή των στρατηγικών για του Ρώμα θα δώσει αποτελέσματα μέσα από επόμενα χρόνια. Οπότε και εμεί βεβαίω ενδιαφέρομαστε εντόνως, να δούμε τι συγκεκριμένα αποτελέσματα θα έχουμε. Αλλά σας τονίζουμε ότι αυτή η ευρωπαϊκή προσέγγιση που την έχουμε εξεργαστεί από κοινό με την ε, κυρία Βίβιαν Ρέντιν είναι κάτι το οποίο είναι μακρόπνο. Δεν ε, οδίδει αποτελέσματα αναγκαστικά ε, κάθε χρόνο. Χρειάζεται μακρόπνοη επένδυση και δεν είναι μόνο ζήτημα χρημάτων. Είναι σημαντικό το ότι αυτή τη στρατηγική την επεξεργαστήκαμε λαμβάνοντας υπόψη τις παλαιότερες ε, δαπάνες όσον αφορά τα άλλα προγράμματα για τους Ρωμά. Επρόκειτο για ενέργειες μόνο από το 2010 με την Task Force. Στη συνέχεια δε, τονίστηκε ότι από τα χρηματοδοτικά μέσα κύριος του Ευρωπαϊκού Ταμείου θα παίξει σημαντικό ρόλο. Αλλά όμως αυτή η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2011 μετά μετετράπησε περισσότερες εθνικές στρατηγικές του 2012. Η δε υλοποίηση των στρατηγικών αυτών βεβαίως απόκειται στις εθνικές κυβερνήσεις και Εξαρτάται επίση η εφαρμογή του από τι ε, δημοτικέ αρχέ, από διάφορε οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών και έχουμε μόνο όλε αυτέ τι δραστηριότητε, τη συνεργασία ε, ε, τα τελευταία χρόνια με, με Δήμου και με αυτέ τι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών. Επίση έχουμε μια σειρά προγραμμάτων στις χώρες, οργανώσει κάποιες άλλες εκδηλώσεις με εμπλοκή των αρμοδίων υπουργών των χρόνων εκείνων, αλλά και με τους δικαιούχους, με προσώπους της Δημοτικής Αρχής. Να τελευταία φορά έγινε κάποια εκδήλωση τον Οκτώβριο στην Ουγγαρία, αλλά πιο πριν στην ε, Βουλγαρία, στο Κόζιτζε της Ανατολικής Σλοβακίας προηγουμένως. Ε, είχε πάει και ο αντιπρόεδρος Επιτροπής, ο κ. Σεφτσοβιτς, και επομένως προέκυψε ε, ότι καταλαβαίνόμαστε με τις αρχές αυτών των χωρών ότι πρόκειται για θέμα προτεραιότητας. Είναι κάτι το οποίο πιέζει. Χρειαζόμαστε υποστήριξη και χρειάζονται υποστήριξη για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Επίσης, ε, οι επαφές με το Συμβουλίο της Ευρώπης, με την Παγκοσμία Τράπεζα και άλλους διεθνείς φορείς, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι εμπλεκόμενοι Όλοι μπορούν να επηρεάσουν τα προγράμματα τα ολοκληρωμένα στην Ανατολική Ευρώπη και δεν μιλώ μόνο για τις νέες χώρες αλλά και για προγράμματα που φτάνουν και έξω από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εκεί χρειάζεται να γίνει συντονισμός κλπ. και ο κύριος Τζορτζ Σόρος με το Ταμείο από την Νορβηγία και αυτός έχει εμπλακεί όσον αφορά το θέμα της κοινωνικής ένταξης των Ρωμά. Πάνω δεν θα λυθεί αυτό το πρόβλημα από τη μια μέρα στην άλλη. Θα έχουμε τα θέματα της απασχόλησης, της παιδείας, της στέγασης. Ε, θα έχουμε αντιμετωπίσουμε και τις δυσμενείς διακρίσεις, όλα αυτά. Ε, είπαμε ότι πρέπει να επιλύσουμε και γι' αυτό σας λέω, πρόκειται για συναρμόδιους περισσότερους επιτρόπους, γι' αυτό σας πω και για τη Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα Και έτσι δεν μπορέσουμε τελικά να έχουμε κάποια αυτά αποτελέσματα. Εάν έτσι επικεντρώσουμε τις προσπαθίες μας. Από όλε τι πλευρές. Επίσης, κάποιοι Ρωμά, το οποίο ισχύει βέβαια για όλους τους Ευρωπαίους, τώρα αυτοί απολάβουν το δικαιώματο της ελευθερίας διακίνηση και θέλουν να το αξιοποιήσουν αυτό το δικαίωμα. Ιδίω εκεί που είναι αφόρητη η κατάσταση στη χώρα της πρόλευσής τους. Ή απλώς θέλουν κάτι το καλύτερο. Υπάρχουν στη χώρα προορισμού κάποιε δυσκολίε, αλλά υπάρχουν και κάποιε προσπάθειε που είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικέ από πλευρά δημοτικών αρχών, ε, περιφερειακών αρχών, όλοι αυτοί αξιοποιούν τα κοινωνικά ταμεία, ούτως ώστε να παρέχουν απασχόληση, παιδεία και στέγαση στους Ρωμά και τι εντοπίζουν τα προβλήματά τους. Προχωρούμε και συνεργαζόμαστε από κοινού και υποστηρίζουμε όποτε χρειαστεί αυτές τις προσπάθειες. Όμως, όμως, θα πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες από τις χώρες που αναφέραμε, εκεί δηλαδή που ε, έχουμε τους περισσότερους Ρωμά, εκεί που ζουν περισσότερο Ρωμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα πολλά έχουμε να κάνουμε όσον αφορά τις αδυναμίες της διοίκησης και έτσι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτές τις ε, περιφέρειες, τις μικροπεριφέρειες ε, να αποκτήσουν κάποια ευημερία εκεί που ζουν δηλαδή οι Ρώμα οπότε και θα έχουμε τότε καλύτερες υλικές συνθήκες για την ένταξη των Ρώμα. Άρα δεν είναι το θέμα ε, του πόσα χρήματα θα ξοδέψουμε αλλά το πώς θα τα ξοδέψουμε προς ποια κατεύθυνση, πώς θα μπορούσουμε τις γενικότερες συνθήκες να τις βελτιώσουμε. Άλλος τομέας τώρα που έχει τονιστεί από τον κύριο Πίπερ ο, το, το πώς κάτι θα γίνει για την ε, απασχόληση, τι θα γίνει με τις ε, εγγύσεις της απασχόλησης των νέων. Πρόκειται για κάτι το οποίο έχει ξεκαθαριστεί. Περισσότεροι εμπλεκόμενοι τώρα αντιλαμβάνονται το ότι δεν πρόκειται για κάποιες εγγύσεις που παρέχονται άμεσα για κάποιες συγκεκριμένες θέσεις Έχουμε τα, τα πρότυπα ε, Αυστρίας και Φιλανδίας και με αυτό το πρόγραμμα θέλουμε να περιορίσουμε την ανεργία των νέων. Δηλαδή αυτοί που είναι κάτω από 25 πραγματικά θα τους ε, πρόσφερε την ευκαιρία ε, κατάρτιση, εκπαίδευση, στάζ, stage τέλο πάντων. Και έτσι δεν θα μένουν ανεργοί όταν τελειώσουν τις σπουδές. Ούτε εδώ είναι θέμα του πόσα χρήματα ξοδεύονται. Είναι το θέμα του πώς θα βελτιώνονται οι δυνατότητες του κρατικού μηχανισμού. Και η προσπάθεια μας εντάθηκαν ιδίως τον Φεβρουάριο στο Συμβούλιο τότε συμφωνήθηκε η υπόθεση αυτή της εγγύησης απασχολής των νέων, αυτή τη σχετική πρωτοβουλία εγκρίθηκε η πρικοδέ των 6 δις και ξεκίνησε μια τέτοια διαδρομή. Να μπορέσουμε να δούμε πώς θα συνεργαστούν όλες οι συνόμοδες αρχές σε όλα τα κρατημέλη και πώς θα αποκτήσουν περισσότερες ε, δυνατότητες, πώς θα χρησιμοποιήσουν τις ε, καλύτερες εμπειρίες που υπάρχουν Γερμανοί, Αυστριακοί, Σουηδοί ε, συνοήθηκαν. Αλλά τώρα όλοι συνεργάζονται και διαμορφώνονται συγκεκριμένε προτάσει, ούτω ώστε να έχουμε τη μεταφορά τη τεχνογνωσία από τι χώρε που ήδη έχουν τέτοια πρότυπα, τέτοια εμπειρία στην εγγύηση για την αποσχόληση των νέων για να μπορέσουν να δανειστούν αυτή την εμπειρία εκεί που τα πράγματα είναι πιο δύσκολα η ακόμα χειρότερα. Χειρότερα τι εννοώ. Εκεί δεν είναι απλή η κατάσταση. Γιατί βέβαια δεν έχουν αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε τα κοινωτικά ταμεία και αναφέρομαι σε κάποιες αδυναμίες, ας πούμε όπως στην Ελλάδα ή στην Ισπανία, που είναι οι χώρες που θα πρέπει κάθε τόσο να ξαναασχολούνται και εμείς μαζί, τι γίνεται με τις αντικανονικότητες, τι γίνεται με το επίπεδο σφάλματος. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλα αυτά θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει αυτή η θετική τάση για την χρήση της εγγύης απασχόλησης των νέων, κάτι το οποίο είναι το θεμέλιο και αφετηρία για πολλές ε, μεταρρυθμίσεις και όσον αφορά τι κρατικέ πίσει απασχόληση, αλλά και όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματικό προσανατολισμό που φέρνει την απασχολησιμότητα ούτω άλλω τέλο πάντων το, κάθε φυσικό πρόσωπο, βρίσκεται κάποια δουλειά κάποια στιγμή. Και υπάρχουν κάποια προγράμματα, σχέδια εφαρμογή, έχουν ε, υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από σχεδόν όλε τι χώρε. Αυτού δηλαδή που, και αυτέ τι χώρε που δικαιούνται να μετέλθουν ε, αυτέ τι εγγύησει. Λειτουργικά προγράμματα είναι αυτά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους του σχετικού καινούριου Ευρωπαϊκού Ταμείου. Ελπίζουμε ότι η στενή συνεργασία των υπηρεσιών της Γενικής Διεθνής για την Επασχόληση και των Κρατών Μελών την άλλη μεριά, συνεργασία αυτή λέγω ότι πρόκειται να ε, ε, ασφαλίσει ότι θα χρησιμοποιηθεί έτσι επιτυχώ το νέο ταμείο, θα έχουμε απορρόφηση, θα χρησιμοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα υπάρχει ποιότητα σε αυτή την πολιτική, στην εφαρμογή της. Και είδαμε σε συναντήσεις στο Παρίσι και στο Βερολίνο και στη Ρώμη, σε συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο. Ε, είχαμε και αρχείους κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέσχουν. Εκεί τα έκανε τις προτεραιότητες και συζητήσαμε τις οικονομικές πτυχές της εφαρμογής της πολιτικής της εγγύησης για την απασχόληση των νέων. Πάντως, σε αυτή τη φάση είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε τους νέους, να ψάχνουν δουλειά. Να ψάχνουν δουλειά, μετά να, να δηλωθούν σε αρμόδιες αρχές και μέσω της συμμετοχής του στο πρόγραμμα θα διαπιστωθεί το πόσο δραστηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα ζητήματα. Φυσικά είναι θεμητό κανεί να αναπτύσσει δραστηριότητα για αυτά. Γιατί έχουμε τι κατευθυντήριε τη απασχόληση που ξεκαθαρίζουν ότι έχει τέτοια εντολή δραστηριοποίηση η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν ώψη τη του 2020 εφαρμόζει κάτι το οποίο δεν θα είναι νεκρό γράμμα, αλλά προκύπτει κάποια δέσμευση όλων των κρατών μελών. Το οποίο μας νομιμοποιεί και ταυτόχρονα μα καθιστά υπευθύνου. Εμάς και τα κρατημέλη. δύναμη των σχετικών διατάξεων της συνθήκης. Έχουμε τη διαδικασία τώρα της οικονομικής διακυβέρνησης και συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό εξάμεινο. με τους σχετικούς μηχανισμούς μπορούμε όλοι αυτούς τους να τους υλοποιήσουμε. Με στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και Κρατών Μέλων. Υπάρχει μια τέτοια αλληλεπίδραση του τι γίνεται σε ε, κοινωνικό επίπεδο και των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης οπότε και εκεί διαδοτρίζονται αυτοί οι στόχοι όπως η ανάπτυξη δυναμικής η εμβάθυνση της ε, ορκιολογικής οδικής αγοράς η οδέ ρυθμός απασχόλησης στα κράτη-μέλη ε, δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα οποία θέλαμε να συμβούν με τη στρατηγική 2020 θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και από πλευρά τη όντω των δύο φύλων και αν θα πρέπει επ' αυτού να να συμβουλεύσουν τα κράτη-μέλη εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και πρόοδου για αυτά. Κυρίως γιατί κάποια από τα σχετικά μέτρα μπορεί να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον το οποίο να ευνοεί την ισότητα των φύλων. Οπότε εδώ πέρα να μπαίνει στο παιχνίδι και το κοινωνικό ταμείο. Ε, ε, I uh, wonder what exactly... Uh, και συνεχίζει ο κύριος Επίτροπος. Θα ήθελα να προσθέσω απλώς πώς... όταν εμείς σημαίνουμε κάποια προβλήματα και τα συζητούμε με τα κράτη-μέλη. Ή τα συζητούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας τονίζω και πάλι ότι προσπαθούμε να εξετάσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Προσπαθούμε να μην γενικεύουμε. Ιδίως όσον αφορά τα πρώτα χρόνια αυτής της σχετικής περίοδου την οποία και συζητούμε, είχαν διατυπωθεί ανησυχίες σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο, όχι μόνο με τις υγείας αλλά και για τον αριθμό υλοποίησης. Όμως, Είχαμε εξαιρετικέ επιδόσεις κατά την τελευταία χρήση, όπως είπα στην εισηγησή μου. Και επομένως, δεν είναι τόσο γενικευμένο το πρόβλημα όσο καμιά φορά εμφανίζεται. Μιλούμε για 65% που εκτανήθηκε για την περίοδο 2007-2013. Το ποσοστό αυτό θεωρείται ικανοποιητικό ρυθμός, άρα έχουμε βελτίωση σε σχέση με το 2008-2009 αλλά μην ξεχνούμε ότι είχαμε τότε τη χειρότερη ύφεση της μεταπολεμικής περίοδου που σίγουρα επηρέασε την εκταμείευση αυτή των πόρων από τα κοινωνικά ταμεία. Άρα επιβαλόταν να γίνει κάποιος αναπρογραμματισμός ε, στη συνέχεια όπως έγινε το 2012 για να δούμε πώς με τον ε, καινούριο προγραμματισμό ε, σε μια σειρά κατών μελών πρέπει να λεφθούν κάποια μέτρα. Πάντως, για το μέλλον θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον κοινωνικό προγραμματισμό, τους ελέγχους, γιατί ο ρυθμός φάλματος εμπόδισε την υλοποίηση. Και όπως και εσείς προγραμματίζεστε για το μέλλον, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μια τέτοια προσέγγιση, αν την προαναφερθήσα πρόκειται, να μας οδηγήσει στο να άρουμε κάποια από τα προβλήματα και αυτές τις αντικανονικέτες που προέρχονται από το α ή β νέο κράτος μέλος. Είναι ο πρώτος τους κύκλους της ε, χρήσης κοινωνικών πόρων τον οποίο τον κλείσανε, τον ξεκινήσαν τέλος πάντων, χωρίς τη σχετική εμπειρία. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί χρήσιμο μάθημα για όλους. Έτσι πάντως εργαζόμαστε στενά με το Κοινοβούλιο και το Ελληνικό Συνέδριο και έτσι θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε στην πρακτική μας. και να βάλουν υπόψη την κτηθή σε αυτήν την εμπειρία και τα σχόλια όλων. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Έχουν ζητήσει εξή τον λόγο. Und dann die Kollegin Gressle, bitte schön. Und der Berichterstatter natürlich. Ja, bitte, Ines. Muchas gracias, presidente. Sí, la señora Andor, siento que he tenido que salir un momento, no he podido estar al comienzo. Συγγνώμη πρόεδρε που δεν ήρθα από την αρχή γιατί είχαμε κάποιους επισκέπτες αλλά άκουσα τα τελικά κατάφερα, ακούσω τους τα περισσότερα πώς ελέγξαν και έχω τις εξής ερωτήσεις. Πρώτα πρώτα. Πέστε μας παρακαλώ τη γνώμη σας κύριε. Τώρα για το 2014, για μας για το 2012. Τι έγινε με τα αποτελέσματα γιατί έχουμε βέβαια τους λογιστικού ελέγχους, αλλά θέλω να δούμε ποια είναι τα, αποτελέσματα όσον αφορά τι δικέ σα αρμοδιότητες. Πέστε μας τη, τη, τη γνώμη σας όσον αφορά το τι αποτελέσματα πετύχαμε με τη χρήση του Γενικού Ταμείου στο επίπεδο της απασχόλησης. Πάει αυτό. Άλλο τώρα. Πώς ελήφθησαν υπόψη τα, τα, τα Γιατί εδώ έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή μας για διάφορα προβλήματα που μας στείλουν την Ισπανία. Το τελευταίο συνέδριο μα έλεγε ότι δεν έγιναν αυτά τα οποία έπρεπε, δεν υλοποιήθηκαν, δεν λήθησαν υπόψη οι προϋποθέσεις. Δηλαδή, δεν εκτελέστηκαν κάποια προγράμματα τα οποία οδηγούσαν σε απασχόληση. Και η Τρόικα πάλι μας επέκρινε. Δεν καταφέραμε επομένω να τηρήσουμε τις ταχθήσεις προϋποθέσεις, μακάρι να είχαμε μπορέσει. Τι να κάνουμε τώρα, πώς θα προσαρμοστούμε στις προϋποθέσεις, στις συνθήκες που επέβαλε η κρίση. Για τις μικροεπιχειρήσεις τώρα. Τι λέτε, ποια θα ήταν τα αποτελέσματα ε, εάν στα σχετικά προγράμματα του 2012 ε, παρέμενε στην γραμμή πλεύσης για τις μικροχρηματοδοτήσεις που αφορούν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γιατί όπως ξέρετε για ΜΜΕ και μικρο ΜΜΕ υπήρξε κάποιο είδους ε, εμπλοκή. Άρα αν δεν γινόταν αυτό, τι συνέπειες θα είχαμε και επιπτώσεις. Πίστη θα με αυτές τις καθαρές δημοσιομικές διορθώσεις γιατί μας μιλήσατε για το πόσο χρειάζεται η επαγγελματική κατάρτιση. Η κατάρτιση τέλο πάντων για τους υπαλλήλου, για τα στελέχη της διοίκησης που θα πρέπει να εφαρμόσουν όπως και οι πολιτικοί τα νέα προγράμματα, τον νέο προγραμματισμό. Για πέστε μας. Εσείς σε ποιο βαθμό φοβάστε ότι η εφαρμογή αυτού του νέου μηχανισμού ε, έγινε στο βάθος και στην πληρότητα που θα έπρεπε. Και έτσι ξεπεράσαμε τον κίνδυνο που συνεπάγεται η μη εκτέλεση των γύρω προγραμμάτων. Η Γκρέσλε. Κύριε ναι, ναι. Επίτροπε, μας παρουσιάσατε μια τεράστια εικόνα των όσων κάνατε, μιλήσατε εδώ πέρα για τους Ρωμά, ε, Νορβηγία, ε, Σόρος, Παγκόσμια Τράπεζα, τα πάντα όλα. Εσεί όμως είστε αυτός με τα περισσότερα κονδύλια. Δεν νομίζω να χρειαζόμαστε όλους τους υπόλοιπου για να κάνουμε κάτι. Για την Παγκόσμια Τράπεζα και το πρόγραμμα με τις ε, μικροπιστώσεις το είχε διαχειριστεί η DG Reggie και τα λεφτά κύριο Σίδε που πήγανε. Άμα είναι δηλαδή να συνεταιριστούμε την Παγκόσμια Τράπεζα. Mm. Δεν το αποκαρήκαμε. Μιλήσατε και στο συνέδριο λήξη ε, τη στρατηγική των Ρωμά, ενός απολογισμού. Ναι. Ας είπατε πως ε, περάσαμε από την κοινή στρατηγική στην εθνική στρατηγική, τώρα πάμε πάλι στου Δήμου, Μα το ζήτημα είναι με ποια πίεση και ποια θέληση για επιτυχία εδώ πέρα κινείται η Κομισιόν. Δεν εφευρέθηκε το 2014 η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. Έτσι, πριν από το 2014 είχαμε πολλούς πολίτες που ήρθαν από άλλες χώρες. Εγώ είδα τα νούμερα από τη Ρουμανία, στη Γερμανία έχουμε 100.000 ανθρώπους που έρχονται το χρόνο. 50.000 από τη Βουλγαρία το χρόνο. Αυτά του 2013 τα νούμερα πριν ε, απελευθερωθεί και για αυτές τις δύο χώρες η διακίνηση. Έχουμε επίσης κάποια επιχειρηματικά μοντέλα ενδιαφέροντα από τη Σλοβακία. Ξεκινάνε οι άνθρωποι για δουλειά να έρθουν να ζητιανέψουν στη Γερμανία. Και η Καθολική και η Ευαγγελική Εκκλησία εκεί πέρα ε, προσπαθούν ε, να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Ε, τι κάνουν. Μένουν 4 με έξι εβδομάδες, έχουν διαπιστώσει οι εκκλησίες, διανυκτερεύουν στο αυτοκίνητο και είναι μπίζνα κανονικά, έρχονται για δουλειά να ζητιανεύσουν. Έτσι. Και οι δήμοι τους οποίους ε, αναφέρεται μένουν αβοήθητοι. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπου στην πατρίδα τους. Το ζήτημα είναι πιεστικό και δεν βοηθάει και τους δήμους τίποτα το να του πω απελάστε τους ή ε, κοιτάξτε αν έχουν μείνει πάνω από τρει μήνε κτλ. Έτσι θα οδηγηθούμε σε, ένα, σε μια χιονοστιβάδα δικών Και είναι αναμενόμενο, έτσι. Δεν, θα, δεν είναι κάτι το οποίο θα προκύψει ενεθρία. Πείτε μου λοιπόν, θα ήθελα, ποια είναι τα τρία πιο επιτυχή έργα για τους Ρωμά. Πείτε μου εσείς. Γιατί εδώ πέρα γυρίζετε από κράτος μέλος σε κράτος μέλος ε, και το πρόβλημα είναι πως ε, από ό,τι φαίνεται υπάρχει και περίπτωση διακρίσεων γιατί σε κάποια κράτη-μέλη δεν θέλουν να δώσουν τα λεφτά στους Ρωμά. Γιατί φοβούνται τους υπόλοιπους. Ε, ούτε αυτό μπορούμε να το επιτρέψουμε έτσι. Είναι ντροπή να υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις. Οπότε, να επανέλθω στα νούμερα του 2012. Έχουμε εδώ πέρα για τη Βουλγαρία Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο απορρόφηση κάτω από 10%. Το είχα πει και στον κύριο Χάν. Και μου απάντησε η Κομισιόν στη σελίδα 42. Και οι ροές των κονδυλίων είναι, είναι πραγματικά σοκαριστικές. Αυτό θεωρώ πως όταν μιλάμε για αυτό το έτος πρέπει να μας πείτε συγκεκριμένα τι κάνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε. Ασχολήθηκε εντατικά με αυτό το θέμα. Πράγματι, είναι δουλειά μας ως Επιτροπή να ρωτήσουμε ποια είναι η αποτελεσματικότητα των ε, κονδυλίων. Και όταν κάποιος δίνει τα λεφτά για τη στρατηγική των Ρωμά, περιμένει και κάποια αποτελέσματα, έτσι. Και βεβαίως ε, θέλουμε, ε, όπως είπα, στο μέλλον ε, σοβαρότερα αποτελέσματα. Και πράγματι αυτό δεν είναι υπόθεση ενός μόνο κράτους μέλους και σε αυτό συμφωνούν νομίζω οι περισσότεροι βουλευτέ ε, και οι περισσότερε κοινοβουλευτικέ ομάδε ότι θέλουμε κάποια αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Πίπερ, ο εισηγητή. Πριν του δώσω όμω το λόγο, θα ήθελα ω πρόεδρο να ρωτήσω το εξή, κύριε Επίτροπε. Έχουμε εδώ πέρα την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, την οποία συζητήσαμε για την αποτελεσματικότητα του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση. Και εκεί πέρα είναι σαφές πως ε, υπάρχουν ε, όντως κάποια άλλα παράπλευρα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν σκοπεύετε εκεί πέρα να επιφέρετε κάποια αλλαγή. Σας ευχαριστώ τώρα. Τον λόγο έχει ο κύριος Πίπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ε, μεταφέρω συχνά τα λόγια του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά θα το κάνω σήμερα. Από μία εφημερίδα. Λέει, έμαθα, ως, ε, σκέφτηκα ως νέος πώς θα φτιάξουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης, αλλά μετά από 20 χρόνια ευρωβουλευτής ε, ε διδάχτηκα πώς θα παραμείνουν τα εθνικά κράτη και καλώς. Ε, αυτό το λέει ο υποψήφιος των σοσιαλιστών. Γιατί ξέρω, πως θα φτιαξουμε τις ηνωμενες πολιτειες ευρωπης αλλα μετα απο 20 χρονια ευρωβουλευτης διδαχτηκα πως θα παραμεινουν τα κάποιους δεσμούς. Αλλά θα ήθελα να πω το εξή. Αυτό το οποίο είπατε για την τοποθέτησή σας ε, για την οικογενειακή πολιτική, για τις συντάξεις, για τους κατώτατους μισθούς, αυτό το οποίο κάνετε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που ορίζεται προϋποθέσεις για ανεξάρτητους επαγγελματίες. Ε, πάρα πολλοί άνθρωποι λένε δεν χρειάζεται να μπλέκει παντού η Ευρώπη, ας ασχοληθεί με κάτι άλλο. Και πράγματι εγώ θεωρώ πως ε, θα μπορούσε να ασχοληθεί με τους περισσότερους ελέγχους εδώ πέρα η γενική σας διεύθυνση. Δεν αναφερθήκατε δυστυχώς στο ζήτημα της αξιοπιστίας των κρατών μελών όμως κύριε Επιτροπέ. Η ίδια η Κομισιόν και αναφέρθηκα στην έκθεση αυτή επανειλημμένως, ανέφερε τις ελλείψεις των κρατών μελών όσον αφορά τις εθνικές ελεγκτικές αρχές και να σας ξαναρωτήσω συγκεκριμένα. Από πού πηγάζει αυτή η αυτοπεποίθηση που έχετε η εμπιστοσύνη ελέγχετε υποθέτω 100% τις δηλώσεις ε, που σας στέλνουν τα κράτη-μέλη για τα επιχειρησιακά προγράμματα, αλλά με ποιο ποσοστό κοιτάτε άμεσα τα ε, προγράμματα μέχρι τον, τελευταίο, μέχρι τον τελικό δικαιούχο. Ή αυτή η εμπιστοσύνη βασίζεται μόνο στις δηλώσεις ε, δαπανών. Δεν είπατε ούτε μία λέξη για αυτό το θέμα. Θέλω να μάθω λοιπόν πώς βλέπετε τις σχέσεις σας έτσι, με τα κράτη-μέλη όσον αφορά ειδικά την αξιοπιστία των δαπανών. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, κοιτάξτε μια που έχει προχωρήσει η ώρα. Παρακαλώ να απαντήσετε, κύριε Επίτροπε, και μετά πρέπει να τελειώσουμε με αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. να ξεκινήσω με τις ε, ερωτήσεις της κυρίας Αγιάλα Σέντερ. Αν δηλαδή έχουμε λάβει υπόψη μας την οικονομική κρίση, να προφανώς ανεφέρθηκα σε πολλές από τις δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει εξαιτία οικονομικής κρίσης, ιδίως όσον αφορά προγράμματα τα οποία είχαμε στην ε, Ελλάδα όσον αφορά τη διαχείριση συγκεκριμένων προγραμμάτων και θα ήθελα επίσης να τονίσω κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ε, πλευρά των προμηθειών όσον αφορά τη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ενίσχυση της ε, απασχόλησης. Κάθε φορά που έχουμε μια οικονομική ύφεση, το βασικό ζήτημα για να διατηρηθεί το επίπεδο απασχόλησης έχει να κάνει με την ζήτηση. Και καταλαβαίνετε ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούμε να ενισχύσουμε τη ζήτηση. Ξέρετε ότι ε, η η ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση είναι αρμοδιότητα οικονομική των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία μπορούν να ελέγξουν άμεσα τα οικονομικά τους δεδομένα. Στα πλαίσια όμως μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης προφανώς έχουμε συντονισμένους κανόνες, αλλά εμείς δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ελέγξουμε ή να επηρεάσουμε το τμήμα της ζήτησης, την πλευρά της ζήτησης και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ δυσχερή συνέπειες όσον αφορά την απασχόληση σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις όσον αφορά τον τομέα της ζήτησης για να εξασφαλίσουμε ότι το εργατικό δυναμικό στα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στον επερχόμενο οικονομικό κύκλο, όταν δηλαδή θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη και όταν θα προκύψει μια νέα οικονομική δραστηριότητα που θα απαιτεί νέες επαγγελματικές δυνατότητες και γνώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να διατηρήσουμε τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και ξέρετε ότι οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερα επιδοτηθεί και ενισχυθεί από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από συγκεκριμένα προγράμματα μικροχρηματοδότησής τους. Ξέρετε ότι κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να έχουμε όσο δυνατόν πιο σφαιρική εικόνα για τις δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη, τις δραστηριότητες ελέγχου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως να συνοψίσει όλες αυτές τις δραστηριότητες σε αυτή τη φάση. Αληθεύει πάντως ότι πολλές φορές έχουμε κάποιες πειραματικές δράσεις, άλλες φορές οι δράσεις αυτές είναι πιο όριμες. Αναφέρομαι σε δράσεις στήριξης των μικρών επιχειρήσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Μερικές φορές βλέπουμε ότι ορισμένες επιχειρήσεις δεν θέλουν να λάβουν κίνδυνο, γιατί ξέρετε ότι ο οικονομικός κίνδυνος ο οποίος πρέπει να καλυφθεί πολλές φορές καλύπτεται από πολλούς διαφορετικούς παρεμβαίνοντες. Καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές πρέπει να γίνει μια κατανομή του κινδύνου σε διάφορους οργανισμούς, πολλές φορές και από τις ίδιες τις κρατικές αρχές. Παρακολουθούμε λοιπόν τον τομέα αυτό και ξέρουμε ότι η επιχειρηματικότητα, το επιχειρήν, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας για την οικονομική ευημερία. Τώρα, η αξιοπιστία των πληροφοριών που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη. Ως προς αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι συνεργαζόμαστε εκ του σύνεγγις με τα κράτη-μέλη που έχουν προφανώς τις δικές τους διαδικασίες ελέγχου και εμείς έχουμε τις δικές μας βέβαια. Και ξέρετε ότι εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό σφάλματος το οποίο σας παρουσιάσαμε. Αντίστοιχο ποσοστό υπάρχει από τα κράτη-μέλη και γενικά τα δύο ποσοστά είναι πάρα πολύ κοντά, τουλάχιστον για τα τρία αυτά τελευταία έτη τα οποία αναλύουμε. Η στενή αυτή λοιπόν συνεργασία με τα κράτη-μέλη και η συνεκτικότητα και ο συντονισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ του συνεδρίου του ελεγκτικού, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των κρατών μελών μα καθησυχάζει και θεωρούμε ότι όντω τα στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη είναι εν γέννη αξιόπιστα. Βέβαια, αν υπάρχουν επιμέρου σημεία τα οποία θέλετε να θίξετε, τότε με ευχαρίστηση εμεί μπορούμε κατά περίπτωση να σα δώσουμε περαιτέρω στοιχεία. Όσον αφορά τώρα τις ερωτήσεις κυρίας Γκρέσλερ για τους Ρωμά. Και πάλι Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε διάφορους παράγοντες όπως ο κύριος Σόρος αλλά και άλλοι οργανισμοί, τους οποίους ανέφερα στην προηγούμενη απάντησή μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνο μία στρατηγική πλαίσιο σε συγκεκριμένο τομέα. Οι εθνικές στρατηγικές από μόνες τους βρίσκονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν αυτές τις εθνικές στρατηγικές, εμείς τις παρακολουθούμε, αξιολογούμε τα αποτελέσματα και όντω υπάρχουν ορισμένε συγκεκριμένε δραστηριότητε, ιδίω στον τομέα τη εκπαίδευση και τη κατάρτιση, που δεν είναι αναγκαστικά επιλέξιμε για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον κοινοτικό προπολογισμό. Στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές προβλέπουμε κάποιους άλλους πόρους και θέλουμε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίσουμε ότι όντως θα έχουμε τις απαραίτητες αυτές δραστηριότητες που θα δημιουργούν τις απαραίτητες ικανότητες για προγράμματα εκπαιδευτικά στις χώρες αυτές. Στις αρχές Απριλίου θα γίνει μια σύνοδος για τους Ρωμά, πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές δηλαδή, και βέβαια είστε ευπρόσδεκτοι να λάβετε χώρα, να συμμετάσχετε σε αυτή την σύνοδο για τους Ρωμά και θα εξετάσουμε διάφορες πτυχές της εφαρμογής διαφόρων στρατηγικών για τους Ρωμά, και θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στο πώς ιεραρχείται, το πώς θέτουμε κατά προτεραιότητα το ζήτημα της εκπαίδευσης όσον αφορά την ένταξη των Ρωμά στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Επ' αυτού λοιπόν θέλουμε να δούμε περαιτέρω πρόοδο, περαιτέρω επενδύσεις και ξέρετε ότι οι επενδύσεις απαιτούν χρόνο προκειμένου να δώσουν τα ευκταία αποτελέσματα. Τώρα όσον αφορά τη δική σας ερώτηση κύριε Πρόεδρε για το EGF, το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Οι αξιολογήσεις που έχουν γίνει προσφάτως, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό Λεκτικό Συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίηση μας έχουν βοηθήσει να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς λειτουργούν τα ταμεία αυτά αλληλεγγύης σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και βλέπουμε ότι ε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι δραστηριότητες ε, EGF έχουν οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, ακόμα και στις χώρες εκείνες που πλήττονται από την οικονομική κρίση και την ύφεση. Πολλές φορές χάρη στα ταμεία αυτά έχουμε δει ότι υπάρχουν ε, πολλοί πολίτες οι οποίοι κατάφεραν να βρουν μια νέα θέση απασχόλησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε είναι ιδιαίτερα θετικά είμαστε πεπισμένοι ότι στη νέα περίοδο προγραμματισμού το EGF θα λάβει υπόψη του όλες αυτές τις διαπιστώσεις των τελευταίων ετών. Θα καταφέρουμε να επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες ακόμα και αν η διαδικασία αυτή είναι εντελώς ξεχωριστή από αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Αποτελεί δηλαδή μια δραστηριότητα εκτός άμεσου κοινωτικού προπολογισμού. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Θέλει ο εισηγητή ξανά τον νου. Όχι. Λοιπόν, σα ευχαριστώ. Κέσονεν, Το λέτε. Ωραία. Ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε. Θα συζητήσουμε οπωσδήποτε ξανά το θέμα και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην Σύνοδο Κορυφή για τους Ρωμά. Πότε θα γίνει, ξέρετε, 6 Φεβρουαρίου. Αν μας στείλετε μία πρόσκληση θα την ε, στείλω στου βουλευτέ, στους αρμόδιους, δηλαδή συντονιστέ των ομάδων. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε τον κύριο Επίτροπο για τι απαντήσει που έδωσε και περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξη. απαλλαγή δηλαδή η απαλλαγή των οργανισμών καλωσορίζω τους εκπροσώπους ε, των αποκεντρωμένων οργανισμών που έχουν ήδη έρθει και χαιρετίζω τον Πέτρη Σάρβαμα, τον εισηγητή και τον Πιέτρο Ρούσο από το ελεγκτικό συνέδριο. Και θα κάνουμε ό,τι και στο παρελθόν. Δηλαδή, θα δώσω τον λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο. Τον λόγο έχει Έχετε λοιπόν το λόγο. Thank you, Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Είμαι ευγνώμων για τη δυνατότητα που μου δίνεται να είμαι παρόν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για να συζητήσουμε την απαλλαγή 2012 για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς με εσά και τους συναδέλφους σας όπως ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα ανάμεσα στον σχετικά χαμηλό οικονομικό κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν αυτοί οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί που συνολικά αντιστοιχούν περίπου στο 1,5% του κοινοτικού προπολογισμού και ανάμεσα στον κίνδυνο που οι οργανισμοί αυτοί αναλαμβάνουν καθότι ασχολούνται με πολύ ευαίσθητες αποστολές και ζητήματα και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι οργανισμοί αυτοί στην κοινή γνώμη. Ας ξεκινήσω με μια σύντομη υπενθύμηση της εντολής του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω την ελεγκτική μας προσέγγιση και τα αποτελέσματα του ελέγχου για το 2012, καθώς επίσης και κάποιες σκέψεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο έλεγχος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου συνδυάζει οικονομικό έλεγχο για την δυνατότητα επίτευξης των ετήσιων οικονομικών δημοσιονομικών λογαριασμών, καθώς επίσης και έναν έλεγχο που αφορά περισσότερο τη συμμόρφωση για την νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών. Στα πλαίσια αυτά το συνέδριο, το ελεγκτικό, προβλέπει μια συγκεκριμένη ετήσια έκθεση για κάθε οργανισμό, η οποία περιλαμβάνει δύο διαφορετικές γνωμοδοτήσεις. Μία γνωμοδότηση για τους λογαριασμούς και μία γνωμοδότηση για τις σχετικές συναλλαγές. Η όλη λοιπόν διαδικασία του ελέγχου μπορεί να οδηγήσει και σε κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την ποιότητα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Το ελεκτικό συνέδριο συνεχίζει να βελτιώνει τους ελέγχους του και στο 2012. Η προσέγγισή μας αναβαθμίστηκε προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη εξοπιστία των ελέγχων και καλύτερε πληροφορίε του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο αριθμό των οργανισμών που υποβάλλονται σε έλεγχο συνεχώ αυξάνεται. Το 2012 ελέγξαμε Κάναμε μάλλον 70 ελεκτικέ αποστολέ με αντίστοιχο αριθμό δηλώσεων αρχικών διαπιστώσεων και το ελεκτικό συνέδριο υπέβαλε 40 ειδικέ αιτήσει εκθέσει που αντιστοιχούν σε 80 γνωμοδοτήσει όσον αφορά του λογαριασμού και την νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών για 40 αποκεντρωμένους οργανισμούς. Για το 2012 λοιπόν η προσέγγισή μας για τον έλεγχο έχει ανανεωθεί τόσο ως προς τη μεθοδολογία όσο και ως προς τον τρόπο υποβολής αναφορών προκειμένου να δίνουμε στο Κοινοβούλιο πιο πλήρες πληροφορίες. Στατιστικές τεχνικές έχουν εισαχθεί πλέον στο όλο σύστημα προκειμένου να μπορούμε να ελέγχουμε μεγαλύτερο δείγμα συναλλαγών. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε υψηλότερο βαθμό αντικειμενικότητας καθώς επίσης και καλύτερη εξοπιστή ελέγχου. Η στατιστική αυτή προσέγγιση συνδυάζεται με μία ανάλυση κινδύνου προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε ένα αντικειμενικό δείγμα το οποίο θα εντοπίσει συγκεκριμένους τομείς κινδύνου. Οι παρατηρήσει τώρα του λεκτικού συνεδρίου υπάγονται σε πέντε συγκεκριμένε κατηγορίε. Αξιοπιστία των λογαριασμών, νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών, εσωτερική έλεγχη, εφαρμογή του προπολογισμού και άλλε παρατηρήσει. Επίση, προβλέπεται και ένα πίνακα συγκριτικό, όπου βλέπουμε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σε σχέση με τις παρελθούσες παρατηρήσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου. Κατά αυτόν τον τρόπο βλέπουμε τι πρόοδος είχε επιτευχθεί από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς όσον αφορά τις παρελθούσε παρατηρήσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου και κατά αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι βοηθούμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει με τη διαδικασία απαλλαγή. Τέλος, αλεξίου σημαντικό, το ελεκτικό συνέδριο έχει προτιμάσει μία σύνοψη των πορισμάτων ελέγχου του 2012 όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς πάντα, που διευκολύνει την οριζόντια ανάλυση των ε, αποτελεσμάτων ελέγχου. Η σύνοψη αυτή, η περίληψη αυτή, εστάλει στους, στις αρχές της για την απαλλαγή και επίσης έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας. Ποια είναι όμως τα βασικά αποτελέσματα, τα βασικά πορίσματα του ελέγχου για το έτος 2012. Το 2012 λοιπόν 40 οργανισμοί, συγκεκριμένα 39 οργανισμοί σύν τον Συνταξιδοτικό Ταμείο της Ευρωπόλ, έχουν ελεγχθεί λοιπόν οι οργανισμοί αυτοί σε σχέση με 39 του 2011 και 32 του 2010. Το Ελεκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και οι 40 οργανισμοί και οι λογαριασμοί τους είναι ιδιαίτερα αξιόπιστοι από κάθε πλευρά. Όσον αφορά τις σχετικές συναλλαγές, έχουν δημοσιοποιηθεί ξεκάθαρες μη τροποποιημένες γνωμοδοτήσεις για, τις, για τους 38 οργανισμούς σε σύνολο 40. Επίσης, μία γνωμοδότηση με συγκεκριμένη αιτιολόγηση ε, εκδόθηκε για τον οργανισμό EIT, για το, Ευρωπαϊ... για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινοτομίας και Τεχνολογίας στη Βουδαπέστη. Δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε συγκεκριμένη χνομοδότηση γιατί δεν υπήρχαν ε, οι... τα απαραίτητα στοιχεία για συγκεκριμένες επιδοτήσεις στον τομέα της έρευνας το 2010. Επίσης, δεν είχαμε τα απαραίτητα στοιχεία όσον αφορά την νομιμότητα και την κανονικότητα των συναλλαγών από την Frontex στη Βαρσοβία. Και γι' αυτό το λόγο στην περίπτωση αυτή το λεκτικό συνέδριο δεν προχώρησε σε γνωμοδότηση γιατί θεώρησε ότι στη διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσματα μπορεί να ήταν αρνητικά. Τώρα, οι μη τροποποιημένε όμως γνωμοδοτήσει για, τις, για του περισσότερου οργανισμού δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αδυναμίες και σφάλματα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι δυναμίες και τα σφάλματα βρίσκονται κάτω από το όριο σημαντικότητας που βρίσκεται στο 2% του προπολογισμού. Χωρίς να θέτουμε να αμφιβόλο την γνωμοδότησή μας, το λεκτικό συνέδριο προχώρησε σε επιπλέον 123 παρατηρήσεις σε διαφορετικούς τομείς που έχουν να κάνουν με όλες τις υπηρεσίες ευρωπαϊκέ, με την εξαίρεση 2. Οι περισσότερες από τις παρατηρήσεις αυτές έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του προπολογισμού και με τους εσωτερικούς ελέγχους. Θα ήθελα να αφαιρθώ τώρα σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Για πολλούς από τους εξωτερικούς αυτούς οργανισμούς, το Λεπτικό Συνέδριο είδε ότι υπήρχε ένας υψηλός βαθμός μεταφορών κονδυλίων, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στο παρελθόν, συγκεκριμένα για το 2012, το Λεπτικό Συνέδριο προσπάθησε να αναλύσει τους λόγους για το υψηλό αυτό ποσοστό μεταφορών και προσπαθήσαμε να αναλύσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα προκειμένου να δούμε αν αυτή η μεταφορά κονδυλίων έχει να κάνει με αδυναμίες στον προγραμματισμό ή αν έχει να κάνει με άλλα εσωτερικά προβλήματα που ενδεχομένω να έχουν οι οργανισμοί αυτοί δεδομένης της πολιτούς φύσης του προγραμματισμού των οργανισμών αυτών. Προσπαθούμε επίση να δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερε πληροφορίε, ιδίω όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση των οργανισμών αυτών. Το λεκτικό Συνέδριο χαιρετήσει την έκθεση προόδου όσον αφορά τον οδικό χάρτη για την κοινή προσέγγιση για τι αποκεντρωμένε αυτέ υπηρεσίε, την οποία δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο 2013. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις κατευθύντριες γραμμές για τον προπολογισμό που θα βασίζεται σε συγκεκριμένες επιδόσεις και προσπαθούμε κατά αυτόν τον τρόπο να ευθυγραμμίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον προπολογισμό και την κατάρτισή του με την ποιότητα της δημοσιονομικής διαχείρισης. Μια άλλη πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η εφαρμογή του νέου δημοσιονομικού πλαισίου, του νέου κανονισμού για το δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από τις αρχές του έτους. Έχουμε εδώ πέρα νέε διατάξει, οι οποίε θα πρέπει να βελτιώσουν την οικονομική δημοσιονομική διαχείριση των υπηρεσιών αυτών. Η έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της κοινή προσέγγισης έχει τονίσει τα αναμενόμενα θετικά στοιχεία από τον συντονισμό των εσωτερικών ελέγχων, καθώς επίσης και από την καλύτερη διαχείριση της πολιετούς φύσης της δραστηριότητας των υπηρεσιών αυτών. Το ελεκτικό συνέδριο χαιρετήσει χαιρετίζει τις νέες αυτές εξελίξεις και θεωρούμε ότι ε, θα πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο τις επιπτώσεις από τον νέο αυτοκανονισμό στα τέλη του 2014. Μια νέα καινοτομία είναι το άρθρο 208 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού που προβλέπει τη χρησιμοποίηση εξωτερικών ανεξάρτητων ελεγκτών και που ε, προβλέπεται ότι θα πρέπει το Λευτικό Συνέδριο να λαμβάνει υπόψη το έργο αυτό των εξωτερικών ελεγκτών. Συζητάμε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις νέες αυτές διατάξεις και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όντως θα δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία για τη διαδικασία ελέγχου των, νέων, των εξωτερικών αυτών υπηρεσιών και ελπίζουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να αποφύγουμε και την επικάλυψη της εργασίας την οποία επιτελούμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και... Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο. Κύριε Ρούσο για αυτή σας την εισήγηση από πλευρά Ελληνικού Συνεδρίου. Κύριε Σαρδόμα Από την κυρία Πρόεδρε, αξιότιμος του Ελληνικού Συνεδρίου, κύριοι Διευθυντές, είναι μεγάλη τιμή μου. Είναι μεγάλη τιμή λοιπόν να είμαι συγκητής για αυτή την διαδικασία απαλλαγής, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά είναι σημαντικό τότε αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα χρήματα των φορολογουμένων. Διότι περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού και ουδενός άλλου. Και επίσης εδώ διακυβεύεται η χρηστή διακυβέρνηση αλλά και η διαφάνεια που διέπουν τις ε, αποκεντρωμένε υπηρεσίε. Θεωρώ ότι θα αξιοποιήσω καλύτερα τον περιορισμένο χρόνο που μου δόθηκε ως εισηγητή, ούτω ώστε να μπορέσω να δω διαφορετικές κατηγορίες και έτσι να θέσω ερωτήματα σε τρεις από τις υπηρεσίες. Τέσσερι, τέσσερι μάλλον, για να μιλήσω. Ε, σε τρεις από τις υπηρεσίες και τέλος το ελληνικό συνέδριο. Θα ήθελα πρώτα πρώτα να ρωτήσω το ERA, το δίκτυο των υπηρεσιών. Μπορείτε να μας πείτε. Απλώς κάτι τη δική σας γνώμη. Τι λέτε για την φετινή απαλλαγή. Για, από πλευρά ε, δική σας, το Ευρωπαϊκό Επίση, το Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία, Να σε σχέση με την ε, νομιμότητα και ε, την κανονικότητα των συναλλαγών. Πέστε μας περισσότερα. Πρέπει να μάθουμε περισσότερα. Περισσότερα και να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι έγινε ακριβώς το 2012 και τι έγινε κατά τις χρήση της προηγούμενης 2011-2010. Ιδίως το 2012. Τότε που ανακαλύψατε ότι σε πολλές περιπτώσεις είχαμε εξάντε επαληθεύσεις λαθασμένες. Πώς ανακαλύψατε αυτά τα λάθη. Πώς αποφασίσατε να έχετε αυτού του είδους τους ελέγχους τους ε, ex post και ακριβώς υπό ποιες συνθήκες αποφάσισε ο οικονομικός ελεγκτής να φύγει από την υπηρεσία σας. Πρέπει επίσης να μας απαντήσετε γιατί φύγατε το 2013 από την θέση του ιστορικού ελεγκτή κατά την Ορσονία το 2012. Επίσης, ο Βαγός Οργανισμός για τα Εξωτερικά Σύνορα, η Frontex. Εδώ υπάρχει ε, η, η ρήτρα εξαίρεση, δηλαδή συνήθως η Frontex δεν χρειάζεται ιδιαίτερου ελέγχου όσον αφορά το τι γίνεται κάποιους ε, δικαιούχου. δεν έχουμε τεκμηρίωση εξάντε πώς εσείς ερμηνεύετε το ότι ο σχετικό κατάλογο ήταν ημιτελή και δεν καλύπτει όλα τα στοιχεία του ενεργητικού. Τρίτον, γιατί υπάρχουν τόσα τροτά σημεία. Επίσης, για τη διαδικασία των προσλήψεων. Όσον αφορά τη διαφάνεια, όσον αφορά την ίση μεταχείριση των υποψηφίων, τι γίνεται σε σχέση με αυτά τα οποία α, απεφάσισε, έκρινε το Ελληνικό Συνέδριο και τέλος. Γιατί δύο τους τρεις διευθυντές έφυγαν από την υπηρεσία σας πέρσι. Πώς επίσης όλα αυτά σχετίζονται με τα προβλήματα τα οποία έχει επισημάνει το 2012 το Ελληνικό Συνέδριο, εάν θεωρείτε βέβαια ότι συνδέονται, σχετίζονται με αυτά τις ε, επισημάνσεις του Ελληνικού Συνεδρίου. Επίσης για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Έχετε εμεί το όσον αφορά την σύγκρουση των ε, κοινωνικών συμφερόντων και θα υπάρξει και πληροφορία στον κόσμο. Πότε θα είναι έτοιμη αυτή η στοσελίδα? Γιατί έχουμε εδώ πέρα κάποια προγράμματα πληροφορική. Ε, Πολλέ φορέ αυτά μπορεί να είναι μεγάλο μπελά, αλλά εσεί σε ποιο σημείο βρίσκεται, πόσο έχετε προχωρήσει όσον αφορά την ε, υλοποίηση αυτή τη βάση δεδομένων. Δεν είναι θέμα 2012, θέμα αυτή τη χρήση. Απλώ αν μα πείτε που βρίσκεστε θα καταλάβουμε καλύτερα σε σχέση με αυτά στα οποία έχει καταλήξει το ελληνικό συνέδριο. Μη μου ξαναπείτε αυτά που είχατε πει το 2011-2012 στις προκαταρκτικές φάσεις. Θέλω να μάθουμε τι ισχύει σήμερα όσον αφορά τις προμήθειες, όσον αφορά αυτά τα προγράμματα τέλο πάντων. Τώρα όσον αφορά αυτή τη μεταφορά, το 79% ε, των πόρων του τρίτου τίτλου. Και μας είπατε ότι έγινε αυτή, αυτή, αυτή η μεταφορά των πόρων έγινε γιατί υπήρχαν ε, ε, κάποιες δαπάσεις που να γίνουν ε, στατηγική σημασία για την πληροφορική. Επομένως, ειδικά για την υπηρεσία ασφαλίσεων και συντάξεων, ΕΙΟΠΑ. τον Δεκέμβριο του 2012 περάφει κάποια σύμβαση, ούτως ώστε να γίνουν αυτού του είδους, αυτού του δηλαδή αυτή τη μεταφορά των σχετικών ποσών του 2013. Και εγώ ρωτώ πώς αυτού του είδους μεταφορά του 79% είναι δυνατόν να γίνεται ε, μόνο σε σχέση με τη μία από άλλες συμβάσεις, γιατί εσείς μας είπατε έχετε μία σειρά συμβάσεων. Πώς αυτές σχετίζονται με αυτή τη μεταφορά αυτού του μεγάλου ποσού και επίσης όσον αφορά τη μεταφορά 2013 προς 2014. Ε, η μεταφορά που θα γίνει λοιπόν το 2013 πάει στο εκπληκτικό 84,5. Πάλι μιλάμε για κάποιο προγράμμα πληροφορική. Για πέστε μας, με αυτές τις μεταφορές, τι, τι, τι, τι θα ωφεληθούμε, τι, θα, τι να ελπίσουμε ότι θα προκύψει. Και τέλος, προς το Ελληνικό Συνέδριο. Έχω μία κάπως πρωτότυπη ερώτηση. Γιατί κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται περισσότερη ομοιομορφία σε σχέση με το πώ το ελληνικό Συνέδριο τη μια χρονιά μετά την άλλη ελέγχει τι υπηρεσίε. Τι θα μπορούσε να γίνει, εάν μπορεί να γίνει κάτι, τι μπορείτε να κάνετε εσεί εις το μέλλον, εάν θεωρήσετε ότι θα επιφέρετε βελτίωση στη διαδικασία της απαλλαγής τι μπορείτε να κάνετε στο μέλλον, τόσο ώστε διαδικασία να περίσει περισσότερη λογική, περισσότερη συνοχή, περισσότερη ομοιομορφία. Γιατί. Σήμερα εγώ τι διαπίστωσα ότι αυτοί που συνοθούνται για να μπουν στην αίθουσα ήταν πάρα πολύ νευρικοί, πάρα πολύ αγχωμένοι, σαν να μην ξέρανε τι τους περιμένει εδώ μέσα. Οπότε τελικά αυτό αντανακλάται σε όλους μας γιατί όλοι μας προσπαθούμε για το καλύτερο. Thank Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή μας για τις παρατηρήσεις που έκανε. Τον λόγο έχει ο Μάσελ Φερσλάιπε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Θα υπογραμμίσω αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος γιατί είχαμε μια συζήτηση μετά την τελευταία διαδικασία της απαλλαγής για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η προετοιμασία της συνεδρίασης αυτής και ελπίζω να βρεθεί μια διαδικασία η οποία θα μας βολέψει όλους. Κύριε Φερσλάιπεν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συγητά, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τον λόγο. Θα επανέλθω. Νομίζω πως αυτό το οποίο είπαν οι κύριοι Ρούσο και Σαβαρμά ήταν πράγματα σημαντικά και καλύφθηκαν εν μέρη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις του εισηγητή. Να πω πως είναι σαφές πως οι υπηρεσίε έχουν δεσμευτεί για υψηλό βαθμό απόδοσης και αποτελεσματικότητας και προχωράμε σε αυτό το μέτωπο. Και βέβαια αυτό ευθυγραμμίζεται πλήρως και με τους στόχους της Επιτροπής σας. Και η διαδικασία της απαλλαγή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία και για εμάς να ξαναδούμε τις βασικές διαδικασίες που σχετίζονται με την διαχείριση των οργανισμών αυτών. Και μπορώ να πω πως έχουμε μάθει αρκετά για το τι απαιτείται από εμάς και πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Γι' αυτό Ακριβώς είχαμε μια πάρα πολύ θετική αξιολόγηση τα τελευταία χρόνια. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο και βέβαια είχαμε και τις παρατηρήσεις που είχαμε που είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας από την πλευρά των υπηρεσιών. Η διαδικασία της απαλλαγής επίσης έχει γίνει πιο διαφανής και χάρη στην εμπλοκή του δικτύου των οργανισμών έχουμε μια καλύτερη ροή πληροφοριών μεταξύ τους και βεβαίως ε, και μία συνέπεια. Νομίζω πως ε, κάποια από τα προβλήματα του παρελθόντος ε, οφείλονται σε παρεξηγήσεις και νομίζω πως η ανταλλαγή πλέον πληροφοριών έχουν έχει παίξει θετικό ρόλο. Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε πώς ε, αναγνωρίζονται πλέον οι οργανισμοί από τα θεσμικά όργανα, ειδικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ελπίζουμε βέβαια αυτό να συνεχιστεί και με τη νέα θητεία του Κοινοβουλίου. Πέρσι τον Ιούνιο η γραμματεία της Επιτροπής σας παρουσίασε τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να γίνει πιο απλή η διαδικασία απαλλαγής ε, και με στόχο ακριβώς να αυξηθεί η διαφάνεια. Και νομίζω πως έχουμε εδώ πέρα ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα του συντονισμού της συνεργασίας και ελπίζω να συνεχιστεί στο μέλλον. Η σημασία του δικτύου που είναι σχετικά πρόσφατο αυξάνεται και βλέπουμε τα ωφέλη όσον αφορά τις καλύτερες επικοινωνίες, και την παροχή συμβουλών οριζόντιας και γενικής φύσης. Ε, και επιμένω σε αυτό γιατί ετέθη το ερώτημα βεβαίως. Τα συγκεκριμένα ζητήματα στην κάθε έκθεση είναι ζήτημα του κάθε οργανισμού ξεχωριστά. Όμως πρέπει να αναφέρουμε πως η πιθανή ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες των διαδικασιών ελέγχου μπορεί να δημιουργήσει έλλειψη συνοχής. Η δημιουργία ενός δικτύου που αφορά με την ανάπτυξη των επιδόσεων και της λειτουργίας είναι κάτι το θετικό για εμάς. Η πρακτική συνεργασία μεταξύ των οργανισμών πλέον είναι πραγματικότητα και πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Και θα συνεχίσουμε βέβαια να ζητούν συνέργειες οι υπηρεσίες. Το ίδιο και στο θέμα των προμηθειών. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων προμηθειών και ο δικός χάρτης προβλέπει πως η Κομισιόν θα στηρίξει τους οργανισμούς αυτούς και έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία να προετοιμάσουμε τυποποιημένες διαδικασίες για να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών και κομισιών. Το πρώτο σχέδιο δε θα είναι στη διάθεσή σας τον επόμενο μήνα και θα το συζητήσουμε. Από την άλλη, είναι σημαντικό να αναφέρουμε κάποια διοικητικά εμπόδια που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας δραστηριότητα. Και εδώ πέρα θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είχαμε πει τον Ιούλιο του 2010. Όλες οι καλές προθέσεις δεν οδήγησαν πάντα στα αποτελέσματα τα οποία ελπίζαμε. Η κοινή προσέγγιση ζητάει απλοποίηση των διαδικασιών ανθρωπίνων πόρων και οικονομικής ε, διαχείρισης, αλλά βλέπουμε πως με το νέο δημοσιονομικό κανονικό κανονισμό πλαίσιο δεν προβλέπεται καμία απλοποίηση. Τέλος, θα ήθελα να υπενθυμίσω την ανάγκη παροχής του ιδίου επίπεδου υπηρεσιών με λιγότερους πόρους, αλλά ξέρετε πως οι οργανισμοί αυτοί ε, σκοπεύουν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους ε, και με μείωση κατά 5% του προσωπικού, όμως ε, για να είναι αυτό δυνατόν και να μπορέσουν να έχουν αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρχει απλοποίηση των συνθήκων εργασίας. Προσεχώς θα υπάρχει και μια νέα διοργανική ομάδα εργασίας, μα δεν είναι όνομα αυτό όμως, με στόχο να εξετάσει την μελλοντική μας ε, χρηματοδότηση. Οπότε και πάλι σκοπεύουμε να εμπλακούμε στο έργο αυτής της νέας επιτροπής ε, για να βρούμε κάποιες βιώσιμες λύσεις. Τέλος, θα ήθελα να προσπαθήσω να δώσω μία απάντηση στο ερώτημα του CT για τα βασικά σημεία τα οποία ανέφερε. Βεβαίως επισήμως θα πρέπει να ζητήσουμε την άποψη όλων των ε, υπηρεσιών, αλλά εάν το δείτε φέτος, νομίζω πως ε, το σημαντικό είναι η εφαρμογή του οδικού χάρτη. Η ενιαία διαφάνεια στους κανόνες και στις διαδικασίες είναι για μας πάρα πολύ σημαντική. Έχω αναφέρει βεβαίως πως ε, συχνά είναι δύσκολο να αντιληφθούμε τις ε, προσδοκίες διαφόρων εταίρων και νομίζω πως η κατάσταση βελτιώνεται. Ακόμα και αν ε, υπάρχουν κάποια προβλήματα, νομίζω πως η σαφήνεια στο μέτωπο αυτό μπορεί να βελτιωθεί ειδικά όσον αφορά τις μεταφορές και το πώς θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε την προβληματική του όλου Οπότε, και βεβαίως το τρίτον είναι το ότι εγώ προσωπικά θεωρώ πως ε, έχει βελτιωθεί η διάθεση συνεργασίας ε, των ε, οργανισμών αυτών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την προσοχή σας. Προσπάθησα να απαντήσω στα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί. Σας ευχαριστώ μιλήσατε ως πρόεδρος του δικτύου των οργανισμών. Τώρα θα ακούσουμε ερωτήσεις, τοποθετήσεις των μελών και θα ήθελα να υπενθυμίσω πως αν ε, θέλετε να απευθύνετε ερώτηση απευθείας σε κάποιο οργανισμό ε, μπορεί να απαντήσει και ο εκπρόσωπός του αν το επιθυμεί. Θα δώσω λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Στάς. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση στην Υπηρεσία Ασφάλειας των Τροφίμων, την ΕΦΣΑ. Παρακολούθησα πάρα πολύ προσοχή και είδα την ερώτηση 30 και την απάντηση που δόθηκε ε, και έχω κάποιες επιπλέον ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Ε, το πρώτο είναι η απάντηση στη σελίδα 67 νομίζω, στη δεύτερη παράγραφο λέει η Εύσα στην απάντηση, στο τέλος παραγράφου, κάποιες ΜΚΟ ζήτησαν η Εύσα να θεωρεί οποιαδήποτε επαφή με τη βιομηχανία ανεξαρτήτως ε, είδους και χρόνου ως ε, συγκρουόμενα συμφέροντα. Ε, για να είμαι ειλικρινής, επειδή ασχολούμαι και με τους NGO και με το παρατηρητήριο της ε, επιχειρηματικής Ευρώπης, δεν έχω δει ποτέ ρητός να απαγορεύουν, να έχουν ζητήσει απαγόρευση ε, των επαφών. Ζήτησαν απλά μία περίοδο πέντε ετών ε, για να μην αναλαμβάνει κανείς θέση μετά από τον δημόσιο οργανισμό σε ιδιωτική εταιρεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει διαβίου απαγόρευση στην συμμετοχή των εργασιών, στη συμμετοχή ε, στις εργασίες ΕΦΣΑ. Δεύτερη ερώτηση, τρίτη παράγραφος. Η τρίτη παράγραφος, ε, τέταρτη πρόταση, παραπέμπεται σε εθνικούς φορείς ελέγχου τροφίμων. Και αυτό το λέτε σαν να είναι κάτι το ουδέτερο. Μα η εθνική ΕΦΕΤ, με συγχωρείτε, είναι μάλλον ο εθνικός αυτός ε, φορέας ε, ο συγκεκριμένος ο οποίος αναφέρεται έχει δημιουργηθεί από την Τανόνε έτσι και στόχο έχει τις δημόσιες σχέσεις με τους δημοσιογράφους και να επηρεάσει την κοινή γνώμη το να παριστάνει έψα ότι δεν υπάρχει εδώ πέρα σύγκρουση συμφερόντων ε, δεν ισχύει αυτό το Εθνικό Ινστιτούτο Τροφίμων δεν είναι τόσο αθώο. Στην ίδια δε παράγραφο παραπέμπουμε πως ε, παραπέμπουμε στην έκθεση του παρατηρητηρίου των επιχειρήσεων που λέει η απλή συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων χωρίς ε, άλλες σχέσεις με τη βιομηχανία για να δώσουν ε, επιστημονικά στοιχεία θα πρέπει να θεωρείται σύγκριση συμφερόντων. Μα, ε, θεωρώ πως πρέπει να παραδεχτούμε αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα το Corporate Europe Observatory είναι πως οι ομιλητές οι οποίοι ε, απασχολούνται σε κάποιους οργανισμούς ε, δεν μπορούν να οργανώνουν τέτοιες ε, διασκέψεις. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να λένε πώς προσφέρουν εμπειρογνωμοσύνη όταν πληρώνονται γι' αυτό νομίζω έχουμε σύγκρουση συμφερόντων. Και μετά η τελευταία παράγραφος σε απάντηση στην ερώτηση 30 δικαίως παραπέμπει η εύσα στο ότι αναζητά μια ισορροπία μεταξύ εμπειρογνωμοσύνης και ανεξαρτησίας για να βρει τους καλύτερους επιστήμονες αλλά νομίζω πως εδώ πέρα δεν αναζητούμε απλά εμπειρογνωμοσύνη εδώ πέρα μιλάμε για κάποια σύσταση πάνελ, εγώ αυτό καταλαβαίνω, το οποίο νομίζω είναι σύγκρουση συμφερόντων. Πρέπει να μην επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων αυτοί οι άνθρωποι. Διαδέλεμε ε, απλά ότι με το να είναι μέλος ενός πάνελ ε, επηρεάζουν βεβαίως. Αυτά, για αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Σαρβάμ, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα απαντήσει μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριος Ντε Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποιες γενικές ερωτήσεις. Αν δει κανείς βεβαίως τον ε, δικό χάρτη της ε, Κομισιόν ε, γίνεται λόγος για αποτελεσματικότητα των ε, οργανισμών αυτών. Κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, λάβαμε κάποιες απαντήσεις, αλλά αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας είναι το αν θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιες εκθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία και για το τι μπορεί να γίνει παραδείγματος χάρη με τη συγχώνευση γραφείων ή και των οργανισμών των ίδιων. Νομίζω κάτι τέτοιο θα μας βοηθούσε. Το δεύτερο είναι κάτι ανάλογο και αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων. Βλέπετε εδώ πέρα στις απαντήσεις πως η ίδια ερώτηση απαντάται με τελείως διαφορετικό τρόπο από τον κάθε οργανισμό. Καλό θα ήταν η Κομισιόν να υποβάλει ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ληφθούν τα μέτρα από τον κάθε οργανισμό, να τα δούμε σε έναν πίνακα για να ξέρουμε το τι γίνεται με την εφαρμογή Υπάρχουν εδώ πέρα κάποια πράγματα τα οποία θέλουν προσοχή, όπως παραδείγματος χάρη αν δούμε τον Άζο και την ε, βέλτιστη πρακτική εκεί πέρα όπου ζητάει παραδείγματος χάρη εθνικούς εμπειρογνώμονες αλλά κάποιοι άλλοι οργανισμοί θεωρούν πως ε, οι εθνικοί εμπειρογνώμονες ε, συμπεριλαμβάνονται στο προσωπικό. Επίσης υπάρχει και το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Δεν ξέρω λοιπόν τι γίνεται εκεί πέρα με την παράταση των ε, συμβάσεων. Θα έπρεπε ίσως οι οργανισμοί να ακολουθήσουν το παράδειγμα της ΕΑΖΑ σύμφωνα με την ε, Κομισιόν το 2013, δηλαδή μετά την ε, ε, περίοδο που κοιτάμε, θα πρέπει να υπάρξει μια προστασία για τυχόν πληροφοριοδότες. Αλλά καλό θα ήταν να μας πούν το τι έχουν κάνει στο μέτωπο αυτό οι οργανισμοί. Και τέλος για την ΕΟΠΑ. Μια ερώτηση. όπου από ό,τι μας λέει η Finance Watch ε, η στην ΕΙΟΠΑ δεν εκπροσωπείται επαρκώς η κοινωνία των ε, πολιτών γιατί βεβαίως θα πρέπει όσοι είναι εκεί να έχουν ε, ε, αρκετή εμπειρία στον τομέα, κάτι το οποίο δεν έχουν βεβαίως συχνά οι οργανισμοί των ενδιαφερομένων. Γιατί η εμπειρία αυτή βεβαίως μπορεί να αποκτηθεί μόνο εντός χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Τι άποψη έχει λοιπόν η ΕΙΟΠΑ εδώ πέρα. Ναι, σας ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Εάν ε, δεν έχει κάποιος άλλος κάποια ερώτηση, περνάμε στις απαντήσεις. Εάν σημείωσα καλά, είχαμε ερωτήσει προς την ΕΦΣΑ, κυρίως από τον Μπαρτ Στάς και ο κύριος Ντε Γιόγκ ε, απευθύνθηκε στην ΕΙΑΖΟ και στην ΕΙΟΠΑ και ίσως και στη Frontex. Ε, ας τα ακούσουμε λοιπόν με τη σειρά ΕΦΣΑ. Η ΕΦΣΑ εκπροσωπείται από τον Dr. Bernard Ουλ, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Θα αναφερθώ καταρχάς στην ερώτηση του κυρίου Στάσα. Σας ευχαριστώ πολύ για το ότι ε, αναφερθήκατε σε ένα πολύ σημαντικό κατεγνώμα ζήτημα, να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην επιστημονική αριστεία και τους ε, χριστούς λογαριασμούς. Εξ αρχής ε, έχουμε πει στην Εύσα ότι χρησιμοποιούμε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Ξέρετε ότι σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εμπειρογνώμονες αυτοί είναι εσωτερικοί. Εμείς έχουμε 1.500 εξωτερικούς εμπειρογνώμονες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βοηθούν την ΕΦΣΑ να εγκρίνει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη συνέχεια για την αξιολόγηση κινδύνου. Να σας δώσω κάποια αριθμητικά δεδομένα επίσης, για να δείτε τι κάνουμε επ' αυτού. Το 2012 αξιολογήσαμε περίπου 7.000, 7.000 ετήσιες δηλώσεις συμφερόντων και ελέγξαμε τις δηλώσεις αυτές σχέση με 33.000 διαφορετικά σημεία που είχαμε σε πολλές συνεδριάσεις τις οποίες κάναμε και αφιερώσαμε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ σε τήσια βάση όσον αφορά το προσωπικό μας και όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι η ΕΦΣΑ αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα της ανεξαρτησίας των εμπειρογνωμόνων πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σοβαρά και όλοι συμφωνούν ε, ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο καθότι από το 2011 και μετά έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε μια νέα πολιτική για να πετύχουμε την σωστή ισορροπία ανάμεσα στην καλύτερη δυνατή εμπειρογνωμοσύνη και στην ε, δυνατότητα να αποφύγουμε οποιαδήποτε εικαζόμενη πραγματική σύγκρουση συμφερόντων. Τώρα κύριε Στάσο, όσον αφορά τις συγκεκριμένε ερωτήσεις σας. Πρώτον, μας είπατε ότι δεν ζητάτε μία επαόριστον απαγόρευση, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όσοι εργάζονται στον συγκεκριμένο αυτό κλάδο, στο βιομηχανικό τομέα, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε πάνελ της ΕΦΣΑ. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι η απασχόληση αυτή μόνιμη αποκλείεται. Δεν υφίσταται το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά το, αυτό το οποίο είπατε, να είναι κανείς ομιλητής ή οργανωτής ή συνοργανωτής επιστημονικού σεμιναρίου, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τον από τη βιομηχανία, από ένα επαγγελματικό κλάδο. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αν η συνδιάσκεψη αυτή βρίσκεται στα πλαίσια έρευνας ενός πάνελ, τότε δεν θα πρέπει να προβλέπετε κάτι τέτοιο. Αν όμως τα αντικείμενα ενδιαφέροντος του, του αυτού είναι εκτός των πάνελ της ΕΦΣΑ, τότε θα πρέπει να επιτρέπεται και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε και εμείς ως ΕΦΣΑ πρόσβαση στους πιο κατερτισμένους επιστήμονες. Και με την πολιτική μας αυτή αποφεύγουμε πραγματικές ή καζόμενες συγκρούσεις συμφερόντων. Αναφερθήκατε επίσης ε, στη συμμετοχή σε ένα Εθνικό Ινστιτούτο Τροφίμων. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και γι' αυτό. Αν μιλάμε για παροχή συμβουλών, επαμοιβή όχι, εμεί δεν κάνουμε κάποια διάκριση, ακόμα και αν δεν υποβάλλεται κάποια πληρωμή για την παροχή αυτή συμβουλών, εφόσον οι συμβουλέ αυτέ εμπίπτουν σε σημείο, σε αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η ΕΦΣΑ, τότε δεν επιτρέπουμε εμεί κάτι τέτοιο. Δεν θα μπορούσε αυτό ο εμπειρογνώμονα ο εξωτερικό να συμμετέχει σε πάνελ τη ΕΦΣΑ, γιατί αυτό αποτελούσε σύγκρουση συμφερόντων. Πάντω νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και λίγο περισσότερο με το ζήτημα τη επιστήμης και τη ανάληψη πρωτοβουλειών και τη διαδικασία λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς για την χρησιμοποίηση εξωτερικών ε, εμπειρογνωμόνων είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μοντέλο και νομίζω ότι αυτό έχει αναγνωρίσει και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τα σωστά επιστημονικά μας αποτελέσματα και πορίσματα. Σαφώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα. Ακούμε πάρα πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία μας λένε μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις ακολουθούμε διάφορες πρωτοβουλίες, θα βελτιώσουμε το σύστημά μας το 2014, είμαστε διαλλακτικοί και ανοιχτοί σε νέες ιδέες και σίγουρα μπορούμε να μάθουμε από όλα αυτά που λένε οι επικριτές μας και κάτι ακόμα να σας πω. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε τόσο πολύ στην επιλογή των υπερογνωμόνων. σαφώ είναι σημαντικό το ζήτημα αυτό και πρέπει να το χειριστούμε σωστά. Ανταυτού νομίζω ότι θα πρέπει να μα απασχολήσει περισσότερο το πόσο ανοιχτή και διαφανή είναι η διαδικασία. Η διαδικασία πρέπει να είναι πιο ανοιχτή, πιο διαφανή, και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να δείξουμε και προ επικριτέ μα ότι εμεί και οι υπερογνώμονέ μα και να του ευχαριστήσω κιόλα επί τη ευκαιρία καθότι κάνουν πάρα πολύ σημαντική δουλειά χωρίς να πληρώνονται. Αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο από την εργασία τους για την πρόθεση της επιστήμης, για την πρόθεση της δημόσιας υγείας, αλλά και αν θέλετε για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μου είπε η γραμματεία πως ο εισηγητής επίσης απίθυνε ερώτηση στον EIT και στο IRA. Μας ακούσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τον εκπρόσωπο της ΕΑΖΑ, ΕΑΖΟ. Κύριε Ντεγιόγκ, σε ποιον απευθυνθήκατε, στην υπηρεσία για το άσυλο ή της αεροπορίας. Κοιτάξτε, είπα ότι η ΕΑΖΑ πρέπει να γίνει παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Είπαμε ότι θα πρέπει και άλλοι να κάνουν τα ίδια, όπως η ΑΖΟ. Καλά. Τότε από πλευρά ΕΑΣΟ έχουμε τον εκδοτικό διευθυντή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που έχετε υποβάλει και όντως να σας απαντήσω όχι τέτοια ευρεία προσέγγιση επιλέξαμε σε σχέση με τη σύγκρουση των συμφερόντων για μία σειρά λόγων. Το έργο το οποίο επιτελούν εδώ πέρα οι μονιμοί υπάλληλοι και οι εμπειρογνώμονες ε, είναι στο δημιουργικό σχήματος. Οπότε είπαμε να μην έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά την σύγκρουση των συμφερόντων. Οπότε και εμεί υιοθετήσαμε αυτήν την λεγόμενη ευρεία προσέγγιση. Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Ο κύριος ε, Χωσέ Μανουέλ Θέτα Γκαρθία από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε, γιατί για την πρώτη φορά που προσερχόμαστε εδώ στην Συμμετική Επιτροπή σας. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να ε, αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω το Συμβούλιο για το 2008 που μαζί με το Συμβούλιο να δώσετε μια ευκαιρία στην ε, καινοτομία με το που συγκροτήσατε την, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο EIT. Βοηθήσατε την επιχειρηματικότητα. Οπότε πέραν αυτή τη ε, εισαγωγής πρέπει να σας πούμε ότι βεβαίω σε όλη αυτή τη διαδρομή μας το 2008, έστειλα στην προσοχή μας το πώς θα σταθούμε στα πόδια μας και είχαμε εγώ το 2011 τον Ιούλιο ε, εργάζομαι εκεί. Τώρα σε σχέση με τα ζητήματα τα οποία ενδιαφέρουν την Επιτροπή σας πρέπει να σας πω ότι από νωρίς καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι το τι θα γίνει με αυτές τις ε, πρικοδοτήσεις τις υποτροφίες και είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας συνεχώς. Από την άλλη μεριά πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή, να έχουμε μια ματιά με κάποιο έλεγχο εξπός τι έγινε στις προηγούμενες χρονιές. Όπως είπε ο εισηγητής, βασικό συμφέρον και ενδιαφέρον εδώ είναι το πώς θα προστατεύσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων, ε, κάτι το οποίο είναι ακόμη πιο σημαντικό ε, στη σημερινή οικονομική συγκυρία θα δείξω δύο ζητήματα τη δική σα ε, αρμοδιότητα. Πρώτα απ' όλα την πρόταση με αυτέ τι υποτροφίε. Θα πρέπει να σα πω ότι επίση έχουμε και πρόοδο όσον αφορά τι κυρώσει κατόπιν ιστορικών οικονομικών ελέγχων. Ε, πάρα πολύ σημαντική η χρήση του 2012 και για τι αλλαγέ και για την πρόοδο, που είπε ο εισηγητή. Σε σχέση με αυτό, θα πρέπει να σα επισύρω την προσοχή στο ότι ε, έχουμε την ιδεολογημένη γνώμη του 2012 του Ελληνικού Συνεδρίου που περιορίζεται μόνο στα όσα έγιναν σε σχέση με τις προτάσεις του 2010. Πολύ σημαντικό αυτό γιατί στην έκθεση του το συνέδριο αναγνωρίζει ότι οι συναλλαγές σε σχέση με το 2011 και τις σχετικές ε, υποτροφίες ε, δεν εμφανίζουν καθόλου λάθη. Οπότε άρα εκ των υστέρων ο έλεγχος είναι πάρα πολύ αξιόπιστος, οπότε άρα ε, το 2010-2011 πήγαμε καλά, το 2011 θεωρηταξεί όπιστο και θεωρείται ότι δεν εμφανίζει λάθη, σφάλματα. Το 2010 επίσης ε, και εκεί είχαμε έλεγχο, οπότε βέβαια ακόμα το 2011 θεωρείται οπιστο και θεωρειται οτι συνέδριο εμείς ακόμα εργαζόμασταν στα τρέχοντα ζητήματα, αλλά πρέπει να σας διαβιώσω γιατί πρέπει πολύ σοβαρά τον έλεγχο του συνεδρίου ότι έχει ολοκληρωθεί ε, αυτή η διαδρομή και τα 2010-2011 όλα έχουν κλείσει τώρα για να ε, δούμε ακριβώς τι θέλει ο εισηγητής, ερωτήσεις του να σας πούμε κάποιες ε, ημερομηνίες σε σχέση με τις υποτροφίες του 2011 με το 2012 τον Οκτώβριο αυτό γιατί υπήρχε μια ιδιορυθμία χρειαζόμαστε ένα χρόνο για να μπορέσουμε με τα κίξ να ένα χρόνο. Και οπότε ε, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε σχέση με αυτές τις υποτροφίες και οι τελικές εκθέσεις ε, δημοσιοποιήθηκαν το Μάρτιο-Απρίλιο 2013, τα ποσά Ιούλιο κατεβλήθησαν και αυτό ήταν ε, αρκετά νωρίς, όσο το λάβει αυτό υπόψη τον το συνέδριο στην έκθεσή του. το για το 2010 πρόεδρε, σημαντικό για το έργο σας. Μάιο 2013 έγιναν οι έλεγχοι και τον ε, Αύγουστο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του και τον Οκτώβριο, Νοέμβριο του 2013 είχαμε τις σχετικές εκθέσεις. Με μεγάλη μας ικανοποίηση μπορούμε να σας πούμε ότι τα χρήματα έχουν ε, ανακτηθεί για τα ΚΙΚΣ. Τώρα, αυτά όσον αφορά την πρόοδο για τις μεγάλες ε, συναλλαγές, το 2012 ειδική εξαιρετική χρονιά, αλλά τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, πιστεύουμε στην αποστολή μας και δεν θέλουμε ε, να ε, συμβεί τίποτα υποτύπων ατυχήματος. Κανένα περιστατικό να μην γίνει ατύχημα. Οπότε βέβαια και τώρα αυτό το οποίο προσδοκούμε είναι το πώς θα συνεχιστεί αυτού του είδους η ακαιρεότητα του Ιδρύματό μας. Τώρα όσον αφορά τη, τα, τις υποτροφίες έκανα την μπορούσα τόσο ώστε να ισχύουν όλα όσα σήμερα σας είπα. Πάντως θέλει ο εισηγητής να μάθει τι κάνουμε όσον αφορά τις ε, κυρώσεις και την αντικατάστασή τους γιατί ήμασταν αρκετά γενναιόδοροι όταν ιδρύθηκε ο οικονομικός για να έχουμε εσωτερική λειτουργία τέτοιου είδους. Όμως απεχώρησε ο προηγούμενο τελικός ελεγκτής, έφυγε από το EIT τελευταία μέρα τη χρονιάς, το 2012. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμεί καθίσαμε σταυρωμένα χέρια γιατί ευθύ αμέσω κάναμε διαγωνισμό, και δεν είχαμε αξιόλογους υποψηφίους, κάναμε ε, ανακοίνωση για δεύτερο διαγωνισμό και το Διευθυντικό Συμβούλιο τον Ιούνιο κατήρθησε μια λίστα υποψηφίων και τελικά ε, προσελήφθη το Σεπτέμβριο του 2013 κάποιος ιστορικός ελεκτής γιατί όπως γνωρίζετε τελικά ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου ενεστώτος έτους. Πέρσι επομένω, κατά κάποιο τρόπο, το δικαιωτικό συνέδριο είπε να φτιάξει μια επιτροπή ιστορικού ελέγχου. Οπότε και έτσι γεφυρώθηκε το κενό μέχρι τότε να αποκτήσουμε ιστορικό ελέγχο καινούριο. Συγκρότησαν αυτή την επιτροπή τον Δεκέμβριο, τότε που μας ειδοποίησε ο ελεγχτή ότι αποχωρεί Θεωρώ ότι ήταν σωστή αυτή η απόφαση να υπάρχει τέτοια επιτροπή. Για πρώτη φορά συγκροτήθηκε τον Μάρτιο. Πάρα πολύ χρήσιμο. Βεβαίω και συμφωνεί η Επιτροπή με το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά την υλοποίηση των συστάσεων. Είναι θέματα διαχείριση και επίση αυτή η, η Επιτροπή κάνει τον ιστορικό έλεγχο και παρέχει τις σχετικές εγγύσεις. Αυτά, Πρόεδρε, και είμαι στη διάθεσή σας για άλλες διευκρινήσεις και ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Frontex κατόπιν. Καλωσορίζω τον κύριο Λάιτινεν, εκτελεστικό διευθυντή της ε, Frontex. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού, απευθύνω επίσης στα μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Όντως, πέντε ερωτήσεις έχουν απευθυνθεί στην Frontex από τον εισηγητή. Θα απαντήσω σε κάθε μία ξεχωριστά. Πρώτη ερώτηση. Έχει να κάνει με το γιατί η Frontex δεν απαιτεί την υποβολή κειμένων για όλες τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τις επιδοτήσεις. Προκειμένου να, απαντή, να απαντήσω με συντομία, θα πρέπει να καταλάβετε ποια είναι η φύση των δράσεων αυτών. Επιδοτήσεις και βοήθεια γίνονται ουσιαστικά στις συνοριακές αρχές των κρατών μελών που χρησιμοποιούν σκάφη καθώς επίσης και αεροπλάνα προκειμένου να καταφέρουν να βοηθήσουν την Frontex και τις ομάδες της καθώς επίσης και τα άλλα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην Frontex να κάνουν την απαραίτητη επιτήρηση. Χρησιμοποιώντας ένα σκάφος ή ένα αεροπλάνο κατά αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να καταγράψουμε όλες τις δαπάνες με τον τρόπο που θα κάναμε για κάποιες άλλες δραστηριότητες. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό αποτελεί αδυναμία και προκειμένου να μετριάσουμε τον σχετικό κίνδυνο, δημιουργήσαμε μία άλλη μορφή συστημάτων, προκειμένου να επαληθεύουμε αν τελικά οι σχετικές αυτές δαπάνες όντως αναλήφθησαν και αν όντως καλύφθηκαν από κοινοτικούς πόρους. Το σύστημα ονομάζεται IEM πρόκειται για τις τρέχοντες, ε, τρέχουσες δαπάνες, τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για την συγκεκριμένη υποδομή που χρησιμοποιείται, για τα συγκεκριμένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται, όπου καταγράφεται κάθε σκάφος, αεροπλάνο ή πλοίο ξεχωριστά και βλέπουμε επίσης ποιο κόστος αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο αυτό μέσο όταν κάνει περιπολίες κάνοντας υπολογισμούς με αυτόν τον τρόπο, καταλήγουμε σε αυτό το οποίο ονομάζουμε patrolling hour, ώρα δηλαδή περιπολίας, κόστος ώρας περιπολίας. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν έχουμε συγκεκριμένη τεκμηρίωση για τη χρησιμοποίηση των στοιχείων αυτών των περιουσιακών, αλλά έχουμε μία κοστολόγηση βάσει της ώρας περιπολίας που κάνουν τα διάφορα αυτά μέσα, στα πλαίσια του νέου αυτού συστήματος που σας ανέλησα. Ένα άλλο σημείο τώρα το οποίο θέλω να αναφέρω και το οποίο είναι λογικό πιστεύω και για μας, είναι να καταλάβουμε ακριβώς ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επιδοτούνται. Ουσιαστικά είναι οι αρχές διαφύλαξης των συνόρων των κρατών μελών. Η φυλακή ουσιαστικά επιδοτείται από τις δραστηριότητες της Frontex, από, την, τον κοινοτικό προπολογισμό. Για τις περιπτώσεις αυτές βέβαια χρειαζόμαστε συγκεκριμένη τεκμηρίωση και γι' αυτό το λόγο σε τήσια βάση περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ αιτιολογούνται μέσω τεκμηρίωσης για τις δραστηριότητες αυτές. Είναι ιδιαίτερα λεπτομερής η τεκμηρίωση αυτή και μπορείτε να τη συμβουλευτείτε μέσω των παραδοσιακών τρόπων και όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμε και άλλα μέσα, άλλους τρόπους και απαιτούμε τεκμηρίωση για όλο και περισσότερους τομείς, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η τρίτη ερώτηση είχε να κάνει με ένα συγκεκριμένο μητρό, το οποίο δεν το είδατε καθόλου στον απολογισμό του 2012. Το 2012 είναι ένα έτος κατά το οποίο είχαμε σημαντικές επιπτώσεις από την Αραβική Άνοιξη που ξεκίνησε το 2011. Το 2011 οι δραστηριότητες της Frontex απέκτησαν και μια άλλη διάσταση. Χρειάστηκε λοιπόν να γίνει μια νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον αφορά τις δραστηριότητές μας, όχι μόνο από επιχειρησιακής πλευράς, αλλά έπρεπε ουσιαστικά να καταφέρουμε να κατανείμουμε και το προσωπικό μας με ένα διαφορετικό τρόπο. Ξέρετε, το διοικητικό μας προσωπικό είναι ιδιαίτερα περιορισμένο. Από την άλλη προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις και ποιος είναι ο κίνδυνος ο οποίος απορρέει από τη νέα αυτή κατάσταση και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ε, μέχρι το 2012 το σύστημα αυτό Μητρώου, το οποίο απαιτείται από τις βέλτιστες πρακτικές, δεν μπορούσε ουσιαστικά να δημιουργηθεί, δεν είχε ολοκληρωθεί. Ποια είναι τώρα τα θετικά νέα που έχουμε. Το Μητρό αυτό πλέον έχει δημιουργηθεί και ακολουθείται και μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για το Μητρό αυτό, που μας επιτρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη σφαιρική εικόνα για το τι διαθέτουμε και τι όχι. Η τρίτη ερώτηση είχε να κάνει με την, το σύστημα πρόσληψης προσωπικού. Στην έκθεση λέγεται ότι υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες και εμπόδια όσον αφορά τη διαδικασία προσλήψεων στη Frontex. Εδώ πρέπει να καταλάβετε ότι έχουμε δύο διαφορετικά τμήματα της διαδικασίας πρόσληψης. Τμήματα που δεν μπορούμε εμείς πολύ εύκολα να προσαρμόσουμε στον τομέα δραστηριοτήτων μας και κυρίως εκεί πέρα όπου έχουμε πραγματικές ένοπλες συγκρούσεις. Ουσιαστικά θέλουμε να δημιουργήσουμε τον απαραίτητο, ένα κατόφλι μάλλον, προσωπικού, να γνωρίζουμε ακριβώς Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ακριβώς στη Βαρσοβία, εκεί που έχουμε την έδρα μας, ποιο είναι το ελάχιστο προσωπικό το οποίο πρέπει να έχουμε, προκειμένου να διοργανώσουμε στη συνέχεια και τις απαραίτητες συνεντεύξεις. Είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε όμως να καταλήξουμε στο ελάχιστο αυτό επίπεδο προσωπικού το οποίο πρέπει να καλυφθεί, ιδίως όταν διεξάγουμε συνεντεύξεις για δύο-τρία άτομα τα οποία υποβάλλουν αίτηση για μια συγκεκριμένη θέση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να θεγραμμιστούμε με τις γενικότερες βέλτιστες πρακτικές. Θέσατε επίσης ένα ερώτημα για το προσωπικό μας, καθώς επίσης και για τους διευθυντές. Έχουμε δύο διευθυντές σε σύνολο τριών, οι οποίοι έχουν φύγει από τη Frontex, όντως. Οι παλιότεροι διευθυντές είχαν μια σύμβαση ορισμένου χρόνου, πέντε ετών συγκεκριμένα. Ενώ ο τρίτος διευθυντής αποφάσισε να υπηρετήσει τη Frontex μέχρι το τέλος της υποεξέτασης περίοδου και ένας άλλος διευθυντής αποφάσει ουσιαστικά να παρατηθεί δύο μήνες αφού του τέθη το ζήτημα ανανέωσης της σύμβασή του. Τώρα, είχαν όλα αυτά κάποιες επιπτώσεις ε, για το 2012. Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρχαν συγκεκριμένε επιπτώσεις. Θα μπορούσε κανείς να πει βέβαια ότι ε, αν είχαμε προσλάβει διαφορετικά άτομα που θα είχαν διαφορετικές επαγγελματικές προτεραιότητες, τότε ενδεχομένω να είχαμε μετριάσει κάπως τα προβλήματα αυτά τα οποία προέκυψαν. Η πέμπτη ερώτηση είχε να κάνει με τις δηλώσεις των προμηθευτών και μας είπατε για ποιο λόγο δεν μπορούμε να έχουμε συγκρίσιμες πληροφορίες από τις διάφορες πηγές που έχουμε από τους διάφορους προμηθευτές μας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι περισσότερες εθνικές αρμόδιες αρχές δεν έχουν ένα κεντρικό σύστημα το οποίο θα μας επέτρεπε να έχουμε μία σφαιρική ισοσκελισμένη εικόνα των πραγμάτων. Πολύ συχνά έχουμε το Υπουργείο Οικονομικών ενό συγκεκριμένου κράτους μέλους, το οποίο παρακολουθεί τους συγκεκριμένους αυτούς ισολογισμούς και πολύ συχνά αναγκαζόμαστε εμεί να απευθυνθούμε στην αρμόδια εθνική αρχή, στο αρμόδιο Υπουργείο και από το ένα Υπουργείο στο άλλο, από τη μία χώρα στην άλλη, λαμβάνουμε και διαφορετικέ απαντήσει. Και τη διαπίστωση αυτή και όλε οι υπόλοιπε διαπιστώσει του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου τι λαμβάνουμε υπόψη μα Πρέπει πάντως να σας πω ότι το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα είναι πολύ δύσκολο για μας, είναι μια πολύ δύσκολη πρόκληση και πραγματικά πολύ φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρουμε εύκολα να τα αποκριθούμε στις προσδοκίες σας που αναλύονται στην έκθεση. Συνοψίζοντας να σας πω ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας όλες τις διαπιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά το 2012 και για το 2013-2014 έχουμε καταφέρει να διορθώσουμε όλα αυτά τα κακό κείμενα. Λειτουργεί ένα νέο σύστημα, όπως σας εξήγησα, και την πρώτη φορά που άκουσα από το ελεκτικό συνέδριο ότι επρόκειτο να προχωρήσει στη μη διατύπωση γνώμης, τότε συνειδητοποίησα πραγματικά και την μεγάλη σοβαρότητα των διαπιστώσεων αυτών που έκανε το ελεκτικό συνέδριο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Λαϊτίνεν. Περνάμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Ο κύριος Κάρλος Μοντάλδο έχει το λόγο, ο κύριος Διευθυντής. Mr. Chairman. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ. Και μας είναι τιμή να προσερχόμεθα και να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία που τη θεωρούμε κορυφαία σημασία. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους από το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά και τους συναδέλφους από τις ε, υπηρεσίες του ιστορικού γνωμελέχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που όλοι αυτοί εδώ παρίστανται γιατί όλοι θέλουμε εδώ να εκτελέσουμε το καθήκον μας για τη λογοδοσία, για την αποτελεσματικότητα και την διαφάνεια. Για να δούμε μία-μία τις ερωτήσεις. Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά τι κάνουμε όσον αφορά ε, το, το, τον ιστότοπο και τη σύγκρουση συμφερόντων θα μπορούσε να είναι η αλήθεια πιο φιλικό στο χρήστη αυτό. Και το είχε χρησιμοποιήσει η προϋπάρξασα επιτροπή που δεν είχε όσους πόρους ε, έχουμε τώρα. Πάντως ε, για την ΕΙΟΠΑ είπαμε ότι θα κάνουμε μια δοκιμή τον Αύγουστο και θα αρχίσει να τρέχει αυτή η υπηρεσία που παρέχουμε από το φθινόπωρο. Όσον αφορά αυτού του κανόνε διοντολογία, κανόνε σύγκρουση συμφερόντων, αυτό το οποίο θέλουμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ευκολία προσβασιμότητα. Α είναι έτσι τα πράγματα. Από τον Ιούνιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τίποτα καινούριο σήμερα απλώ. Δεν τα έχουμε όλα αυτά βάλει στη θέση του, δεν τα έχουμε ε, τοποθετήσει ούτω ή στο website. Το πρώτο το οποίο θέλουμε πάντως να προσφέρουμε είναι την προσβασιμότητα. Να μπορεί κανείς να μπει εκεί για να μπαίνει εκεί εύκολα. Έχουμε τους επόπτες, έχουμε το διοικητικό συνέδριο, ήδη αυτά έχουν ανέβει στο website. Την αρχή διαχείρισης της ΕΙΟΠΑ και φέτος είχαμε μία δυσάρεστη κατάσταση. Ένας από τους συναδέλφους, γιατί πριν είχαμε όλες τις πληροφορίες στο website, τις πληροφορίες και τα τηλέφωνα, ε, απειλήθηκε. Απειλήθηκε, ε, κάποιος του είπε ότι θα αυτοκτονήσει, του να σε από την γερμανική αστυνομία και αποφασίσαμε ότι θα έχουν περισσότερες πληροφορίες, κυρίως ε, το χειριστικό όργανο και οπότε είχαμε τους κανόνες που εγκρίθηκαν για σύγκρουση συμφερόντων για το υπάρχον προσωπικό και για το Συμβούλιο των Εποπτών και εγώ ως εκτελικός διευθυντής ήμουνα αυτός ο οποίος υπέραψε τους διορισμούς αλλά δεν έχω διορίσει όλα τα μέλη του Συμβουλίου οπότε έχουμε ε, ε, τη μνήμα όλων αυτών στο website. Έχουμε και κάποια κώδικα διοντολογία, τον οποίο ακολουθούμε, ε, διαφάνεια και ε, διοντολογία, ισχύουν από την αρχή. Εγώ ήμουν ο υπάλληλο ο αρμόδιος για τη φορμή της διοντολογίας, για τη χρηματοδότηση, για τις συμβατικές σχέσεις με τους εταίρους μας, ε, και τις οικογένειές τους, τι θα πρέπει να πληρούν όσοι υπηρετούν εκεί στην ΕΙΟΠΑ και είπαμε ότι θα πρέπει να κάνει κάποιος τέλο πάντων κάποιες κινήσεις, να εκτελεί κάποια διαδικασία όταν θέλει να εργάζεται στην ΕΙΟΠΑ. Τελευταίο, αλλά σημαντικό, είναι κάτι το οποίο πρόσφατα εγκρίναμε, είναι κάποια πολιτική πώς επιτελούμε τις λειτουργίες μας ε, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να δούμε ε, πού υπάρχουν οι κίνδυνοι για τη λειτουργία της υπηρεσίας. Έχουμε έρθει σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτή την καταγραφή των κινδύνων. Και με τους ε, επόπτες ε, συμφωνήσαμε. Επίσης έχουμε αυτό το πρόγραμμα πολιετούς χαρακτήρα 2003-2015. Τα πράγματα είναι απλά για αυτό το πρόγραμμα και τα καλά μαντάτα ότι αυτό το πρόγραμμα εξαρτάται από ένα μεγαλύτερο που λέγεται Solvency 2. Φενικιώτα 2. Ε, τρέχει υπό τον έλεγχο του, και του Κοινοβουλίου εδώ και 13 χρόνια και δόθηκε το πράσινο φως για αυτό το πρόγραμμα, οπότε ξέρουμε ότι θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2016 το 2014 και το 2016 θα πρέπει να αναλυθούν και συνέργειες ούτως ώστε το 2016 να γίνει υποσαρμογή αυτού του προγράμματος στην, ε, και τους κανόνες εποπτείας σε σχέση με τους κινδύνους. Να πως έχουν τα πράγματα σήμερα και είναι σαφές ότι μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2014 θα πρέπει να έχουμε αναπτύξει προτυποποίηση και συλλογή στοιχείων ούτως ώστε το 2015 όλα αυτά να μπορούν να ελεγχθούν και να χρησιμοποιηθούν. 2014 για προτυποποίηση και τα δεδομένα με αυτήν την που λέγεται ταξόνομη, συγγνώμη. Σας, δεν είμαι ειδικό σε αυτά, Ίσως τα αναφέρω όπως τα ξέρω. Και θα πρέπει στις εθνικές ευρωπαϊκές υπηρεσίες και σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείε που θα υπαχθούν σε αυτό το Solvency 2 να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει με τα δεδομένα σε κάποιο φύλλο Excel και θα έχουμε αυτό με τη μετάφραση όποτε χρειάζεται και όσον αφορά τώρα τις εθνικές ευρωπαϊκές αρχές θα τους δώσουμε ένα toolkit για αυτού του είδους τα δεδομένα και το τελευταίο στοιχείο είναι μια κεντρική βάση δεδομένων και έτσι θα βοηθούν όλοι όσοι δεν είναι ειδικοί όπως δεν είμαι εγώ για να μπορούν να δουλέψουν όλες αυτές τις εταιρείες. Άρα σημειώνεται πρόοδος και επομένως πρώτη από το 2015 θα έχουμε ό,τι χρειάζεται για να τρέξει το Solvency 2. Τι ποσόν σημαίνουν όλα αυτά. Όσον αφορά τις λύσεις της πληροφορικής, για αυτό το πρόγραμμα 2015 είπαμε ότι θα είναι 8,4 εκατομμύρια. Όταν αφορά την υποδομή και την αρχιτεκτονική της πληροφορίας είναι 5,4 εκατομμύρια ευρώ. Άρα συνολικά μιλούμε για ένα τεράστιο πρόγραμμα όσον αφορά τον προβολισμό που φτάνει στην πληροδότηση των 14,8 περίπου εκατομμύρια. Κάτι άλλο το οποίο ρώτησε ο συγητής έχει σχέση με τις μεγάλες σημαντικές μεταφορές. Είναι το 2012 και κατόπιν πήγαμε το 2013. Βέβαια το 2012 έχουμε τη διαδικασία απαλλαγή που έγινε, αλλά γι' αυτό και είπαμε στο Κοινοβούλιο ότι επίση θα ήταν σημαντικό <clears throat> να τα εντάξουμε αυτά στο ίδιο πλαίσιο και άρα η ερώτηση είναι αυτό το 79% πώς σχετίζεται με αυτά τα προγράμματα της πληροφορικής όχι, δεν σχετιστεί. Έχουμε 2,2 εκατομμύρια και άλλους τέσσερις τομείς που έχουμε μεταφορες μεταφορές. όλα έχουμε μια κοινή σύμβαση που την αναλάβαμε με την ε, ΕΣΜΑ που είναι η ασφάλεια των δικτύων. ΕΣΜΑ. Και έχουμε επίσης Έχουμε κάποια μέλη εδώ που είναι δύο υπηρεσίε και σε εμά και, στην... και, εκεί. Και οπότε ε, τελικά διπλασιάστηκε το κόστος και μιλούμε για 193.000 ευρώ. Με τις εποπτικές αρχές έχουμε 30 εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, πάρα πολύ φιλοδοξό πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα αυτό έχει να κάνει και με κάποιες πρωτοβουλίες για σεμινάρια του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου. Αλλά κατόπιν το 2012 και το 2013 αποφάσισαν οι επόπτες μια που είχαν κάποια από τα μέλη μας σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, αποφάσισαν ότι de facto χρειάζονται περισσότερη κατάρτιση και άρα θα έπρεπε να γίνει περισσότερη οικονομική υποστήριξη. Και επομένως αυτό δημιούργησε πρόβλημα όσον αφορά την δέουσα δικαιολόγηση και είπαμε ότι θα πρέπει να έρθουν στην ε, διάφοροι εθνικοί ελεγκτές στην κατάρτισή μας, άλλες 40.000 ευρώ, ενταλή πληροφοριών, 49.000 ευρώ και άλλες 60.000 όσον αφορά άλλα προγράμματα πληροφορικής. Άρα, αν τα αφήσετε όλα αυτά για το κοινή σύμβαση, την κατάρτιση των εποπτών, πάμε σε περίπου 100.000 ευρώ. Φτάνουμε το 2013 και εκεί για 85% ε, ποσοστό το οποίο θα πρέπει να μεταφερθεί. Και ε, ήδη με το που τα λέμε αυτά ε, δουλεύουμε με διαφάνεια και υπάρχει και άλλο πρόγραμμα πληροφορικής, πάρα πολύ σημαντικό, το 2012 είχαμε συνολικά 2,8 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τις δύο φάσεις αυτού του προγράμματος πληροφορικής Πάμε στα 3,8 εκατομμύρια το 2013 και από αυτά καταβάλαμε το 6% και τα υπόλοιπα πρόκειται να καταβληθούν κατά το 2013. Όχι, συγγνώμη, 14 λέει ο Και το υπάρχει και κάτι τελευταίο που πρέπει να σας αναφέρουμε, είναι ότι πολλές φορές πρέπει να αναφέρουμε τη μεταφορά όταν δεν συνδέεται με κάποιο πρόγραμμα. Και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι εδώ πέρα έχουμε αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη σύμβαση πλαίσιο και από αυτό το 79% που μεταφέρει από το 2012 έχουν εκτελεστεί πάνω από τα 99% αυτού. Αυτό αφορά την τρίτη ερώτηση του συγητή και η τελευταία ερώτηση του συγητή έχει να κάνει με την ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΕΙΟΠΑ. Μπορώ να σας πω για το ΕΙΟΠΑ, αλλά μπορώ να σας πω και για τους συναντούς των άλλων υπηρεσιών. Έχουμε ιστορικές τέτοιες ομάδες από τους δικούς μας ε, ειδικού και αυτούς που προέρχονται από τις εθνικές ευρωπαϊκές αρχές. Οπότε έχουμε και αυτές τις ομάδες των εμπλεκομένων και ωφελούμεθα από την συμμετοχή αυτών των ε, τρίτων. Είτε είναι πανεπιστημιακοί, βιομηχανία, συνδικαλιστές κλπ. Οπότε είναι σωστό να αναφέρουμε ότι η πρώτη διαδικασία επιλογής θα επιδεχόταν βελτιώσεις που έγινε το 2010. Η υπηρεσία μας όμως τότε δεν είχε ακόμα συγκροτηθεί και επί τη βάση του κανονισμού πρέπει να διαβάσετε γιατί καμιά φορά δεν είναι τόσο ξεκάθαρο πώς εφαρμόζονται σχετικά κριτήρια πρώτα-πρώτα από τις προηγούμενες πρακτικές της προϋπαρχούσης επιτροπής. Οπότε και γι' αυτό και αρχίσαμε να επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις. Ε, συνοηθήκαμε με τον διαμεσολαβητή, να δούμε αυτούς που είχαν ήδη υπηρετήσει τι, τι θα μπορεί να γίνει. Κάναμε κάποιου κανόνες επιλογής οι οποίοι εφαρμόστηκαν πέρσι το καλοκαίρι και οπότε κατά τη γνώμη μας ε, έτσι καλύπτουμε και ο Σεστατο Finance Watch και ο Ombudsman. Οπότε έτσι θα καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή επιλογή για το stakeholder group. Τώρα, πρώτα πρώτα υπάρχει εδώ πέρα μια ανισορροπία και συμφωνώ μαζί σας Δυστυχώς συνέβη και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Αλλά λέει ο οργανισμός ότι 10, 10 από τους 30 πρέπει να προέρχονται από τη βιομηχανία. 5 θα πρέπει να προέρχονται από ανεξάρτητα πανεπιστήμια. Αυτή είναι δύο περιορισμοί. Και κατόπιν έχουμε άλλες 6 κατηγορίες που αναφέρονται και θα πρέπει να ισχύσουν. Και έχουμε εδώ πέρα 5 πανεπιστημιακούς, σαν παράδειγμα, και έχουμε τη σωστή ισορροπία όσον αφορά τη, την προέλευση, γυναίκες άντρες κλπ. Από τους από ασφαλιστές έχουμε έξι αιτήσει για τις πέντε θέσεις, αλλά προέρχονται από το ίδιο κρατός μέλος κατά σύμπτωση. Άρα τι θα κάνουμε, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το, το ελάχιστο που επιβάλλεται όπως κάνουμε τους τρεις, γιατί αλλιώς θα κατηγορηθούμε για δυσμενή διάκριση από τη βάση εθνικότητας ή τι θα κάνουμε, ή θα πούμε δεν κάνουμε τίποτα γιατί θα πάνε αρκετά καλά. Άρα έγινε μια διαδικασία, ε, θεωρήθηκε αξιόλογη, τη συζητήσαμε τον Ombudsman, η κατάσταση είναι αρκετά καλή όσον αφορά τι μας λένε ενδιαφερόμενοι, αλλά πολλές φορές στην πράξη τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και τελικά η πρόεδρος ε, είναι γυναίκα και είναι, ε, από την ομάδα των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ για την ε, εκδομένη απάντησή σας κατά το οποίο δείχνει βεβαίως πως σας απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα. Δύο ακόμα οργανισμούς περιμένουμε και η Κομισιόν οπωσδήποτε θέλει το λόγο. Οπότε θα δώσω τον λόγο απευθείας στην ΕΑΖΑ. Ο κύριος James Wood, μόνιμος ε, γραμματέας για το συντονισμό των οργανισμών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διοικητικά υπάγομαι στην ΕΑΖΑ. Οπότε ευχαριστώ που δώσατε τον λόγο στην ΕΑΖΑ. Η ΕΑΖΑ δεν έχει σχόλια ή δηλώσεις και δεν έχω να κάνω και καμία δήλωση γιατί βεβαίω εργάζομαι για τον πρόεδρο του δικτύου, τον κύριο Φερσλέπ, εδώ εξεφωνήμων, οπότε έχει ήδη απαντήσει ο ίδιος ο πρόεδρος. Μάλιστα. Έχουμε τι έχουμε ακόμα, την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων. Mm, ναι. Μου αν θα θέλατε να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ. Ε, λειτουργεί το μικρόφωνο, ναι. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες για την συζήτηση, αλλά σημαντικό είναι τώρα βεβαίως να ακούσουμε την Κομισιόν. Και βεβαίως να δούμε πως δημοσιεύσαμε την έκθεση ε, δραστηριοτήτων για την κοινή προσέγγιση, το τι έχουμε κάνει το 2013 και στην έκθεση αυτή βεβαίω σημαντικό κομμάτι είναι η δράση 34, ο περίφημος οδικός χάρτης ε, για το τι γίνεται με τα συγκρόμενα συμφέροντα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί διακούστηκαν πολλά, αλλά ξέρετε πως η Κομισιόν τον Δεκέμβριο που μας πέρασε δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη και διαχείριση συγκρουόμενων συμφερόντων στις υπηρεσίες μας. Και γνωρίζετε πως γίνεται κάποια δουλειά, δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες γιατί υπάρχουν κάποιοι τομείς που αναφέρονται, αλλά η δουλειά συνεχίζεται. Αυτό σημαίνει πως θα συνεχίσουμε και φέτος και σε πιο ακριβείς ε, κανόνες με βάση τις κατευθύνες γραμμές κομισιών. Θεωρώ λοιπόν πως εδώ πέρα υπάρχει αρκετή πρόοδος και εξελίξεις και χαιρόμαστε για την εξέλιξη του οδικού χάρτη και νομίζω πως είναι αποτέλεσμα και της ε, διοργανικής ομάδας εργασίας. Το ότι δηλαδή είχαμε πλέον σαφείς κατευθυντήριες γραμμές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Φεσλάιπεν από την Κομισιόν. Δεν θέλει το λόγο. Τελειώνουμε λοιπόν με το ελεγκτικό συνέδριο και μετά με τον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Σάρβαμα για τη σημαντική αυτή ερώτηση που νομίζω πως πάει κατευθείαν στο κορυφαίο θέμα που μας απασχολεί κατόπιν. Αν κατάλαβα καλά το ερώτημα του κυρίου Σαβάρμα ζήτησε μια πιο συνεκτική αντιμετώπιση από το ελεγκτικό συνέδριο γιατί θεωρεί πως ε, ε, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των οργανισμών. Όντως, όντως αυτό ισχύει γιατί γιατί κάποιες από αυτές έχουν ρυθμιστικές εξουσίες, ε, άλλες είναι παρατηρητήρια, άλλες πάλι ε, κάνουν έρευνα. έχουν ε, διαφορετική οργάνωση, μέγεθος και ε, διοίκηση, διοικητική δομή. Αν κατάλαβα καλά λοιπόν το ερώτημα του κυρίου Σάρβαμα, από ό,τι φαίνεται ε, θα έπρεπε να υπάρχουν πιο ενιαία κριτήρια και να λαμβάνετε υπόψη με αυτή η διαφορά. Γιατί, εάν πάλι κατάλαβα σωστά, ακόμα και αν φαίνεται περίεργο, η συνεκτικότητα θα προέλθει μέσα από την ε, διαφορά που υπάρχει. Θα ήθελα να πω πως ο έλεγχος όπως προβλέπεται στην συνθήκη και στον δημοσιονομικό κανονισμό και στον κανονισμό πλαίσιο, διαφέρει. Γιατί ε, μιλάει για 100% έλεγχο κανονικότητας και νομιμότητας. Οπότε ε, είναι πράγματι ενιαίος, αλλά υπό μία άλλη ενιαία. Δηλαδή, πρέπει να ελέγξουμε για κάθε ε, υπηρεσία, τους λογαριασμούς, ε, το εάν υπάρχουν και το εάν οι συναλλαγές είναι νόμιμες και κανονικές. Και στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να λάβουμε υπόψη τη αφορά μεγέθους, αποστολής κτλ. Γιατί οι κανόνες ε, ορίζονται από τον νόμο. Παρ' όλα αυτά γνωρίζω πλήρως την ανάγκη που έχει το Κοινοβούλιο και ο εισηγητής να έχουν αυτές τις πληροφορίες. Βεβαίω αυτές τις πληροφορίες ε, πρέπει να δίνονται πρώτα απ' όλα από το ελεγκτικό συνέδριο στις ε, εκθέσεις του, αν μπορεί να δίνει τις απαντήσεις κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί έχουμε λίγους πόρους Ε, τα κάναμε αυτά πρόσφατα και ελπίζουμε να δοθεί και μια συνέχεια, αλλά ε, ήδη ευθύς εξ αρχής από όταν αναλάβαμε αυτή την ευθύνη προσπαθήσαμε να διευρύνουμε το πεδίο του ελέγχου που επαναλαμβάνω ξανά πως πρέπει να αφορά την ομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών και να βρεθεί η σύνδεση μεταξύ διαχείρισης του προπολογισμού και της διοίκησης καθεαυτής. Και λέγοντας κατά περίπτωση, παραδείγματος χάρη, τι γίνεται με τη μεταφορά κοντιλίων από έτος σε έτος, αν υπάρχουν ε, υπερβολές ε, στις μεταφορές, αν ε, αυτό οφείλεται σε έλλειψη ή λάθος σχεδιασμού ήταν πολυετής η δραστηριότητα και το απαιτούσα. Το ίδιο και για υπερβολικές ακυρώσεις. Ε, ε, ε, της χρηματοδότηση, κάτι το οποίο θεωρητικά θα μπορούσε να σημαίνει, παραδείγματο χάρη, το ότι η χρηματοδότηση που δίνεται από την Κομισιόν είναι υπερβολική σε σχέση με τα καθήκοντα του οργανισμού. Ε, για να καταλήξω λοιπόν. Ναι, να ληφθεί υπόψη η διαφορά Κάτι το οποίο βέβαια αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο. Κάτι το οποίο θα πρέπει να μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε μια συνεκτική εικόνα, υπ' αυτή την έννοια βεβαίως που προανέφερα. Αλλά κάπου εκεί σταματάει η δική μας η αρμοδιότητα και τα συμπεράσματα είναι η δουλειά του Κοινοβουλίου. Επαναλαμβάνω πως προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε με τα μέσα που έχουμε για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ρούσο, τον λόγο τώρα έχει ο εισηγητής. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω θερμότατα όλους σας που απαντήσατε σε ερωτήσεις μου. Αυτό πραγματικά καταδεικνύει ότι δεσμεύεστε πραγματικά να τα αποκριθείτε στα καθήκοντά σας, αυτά για τα οποία σας επέλεξαν. Βέβαια, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ε, ακόμα πρέπει να γίνουν σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουμε σε αυτόν τον ιδανικό κόσμο που θέλουμε να καταλήξουμε. Δεν έχουμε φτάσει όμως ακόμα εκεί. Ας συνεχίσουμε όμως το δρόμο αυτό των βελτιώσεων και των διορθώσεων. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Στην περίπτωση της Frontex, νομίζω τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Τα πράγματα δεν είναι απόλυτα, δεν είναι άσπρο μαύρο. Και σίγουρα η απαλλαγή αυτή δεν θα πρέπει να κινηθεί σε αυτό το πνεύμα. Ακούγοντας λοιπόν τον εκτελεστικό διευθυντή της Frontex, ο οποίος έδωσε πλήρεις απαντήσεις, Σκέφτηκα λοιπόν ότι ενδεχομένως να ζούμε σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Με άλλα λόγια, αυτά τα οποία μας λέει με απόλυτη συνεκτικότητα το λεκτικό συνέδριο όσον αφορά την νομιμότητα και την κανονικότητα των λογαριασμών, διαφέρουν πάρα πολύ, ανήκουν σε ένα διαφορετικό κόσμο από αυτόν μέσα στον οποίο λειτουργεί η Frontex ενδεχομένως να βρίσκεστε σε μια κάποια άλλη διαφορετική διάσταση. Αυτό το οποίο θέλω να πω ουσιαστικά είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου οι δύο αυτοί φορείς να έρθουν πιο κοντά, να καταλήξετε να μιλάτε την ίδια γλώσσα με το λεπτικό συνέδριο και θα γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Μου δόθηκε εντύπωση ακούγοντά σα ότι ενδεχομένω τα μέσα τα οποία χρησιμοποιείτε, ο παραδοσιακός τρόπος που χρησιμοποιείτε για την απαλλαγή και τον έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αποκρίνονται πάντα στις ανάγκες που εμείς οι ίδιοι τελικά προσπαθούμε να καλύψουμε μέσω των οργανισμών μας. Ενδεχομένως να γίνεται κάπως φιλοσοφική η συζήτηση, αλλά βλέπετε ότι ως ε, εισηγητής ε, για την απαλλαγή των οργανισμών τα πράγματα σίγουρα δεν είναι εύκολα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά θερμότατα για την συμμετοχή σας. Βλέπω ότι έχετε λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη σας όλο αυτό εγχείρημα και πιστεύω ότι μέσω της ακρόασης αυτής καταφέραμε να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση και σίγουρα θα καταφέρουμε με μεγαλύτερη ευκολία να επιτελέσουμε το μέλλον μας στο έργο. Πρόεδρος, ε, σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι για την ε, έκθεση αυτή. Τον εισηγητή ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση την οποία κάναμε. Ολοκληρώνεται η δημόσια συζήτηση και ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό και θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας αύριο το πρωί, τη συνεδρίαση.